surely, surely we were on our way to the exchange of views on this second. Έχουμε λοιπόν την ανταλλαγή απόψεων ε, ε, σχετικά με τη δεύτερη έκθεση υποπτία τη κοινή αρχή ελέγχου του Ευρωπόλ. Τη Ευρωπόλ μάλλον. Και μια και θέλουμε διαφάνεια σε, αυτά τα, σε αυτό το κοινό εποπτικό σώμα. Έχουμε και δημοσίως ε, την έκθεση αυτή με τις ε, βασικές παρατηρήσεις. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ράινχαρτ Πρίμπε, που είναι Διευθυντής Εσωτερικής Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών, που θα μας μιλήσει για την ε, επερχόμενη αναθεώρηση ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτείων για το TFTP. Και έχουμε επίσης μαζί μας την κυρία Ιζαμπέλ Κρούς, που είναι πρόεδρος του κοινού εποπτικού σώματος, GSP της Europol, που θα μας κάνει μια παρουσίαση των πορισμάτων της δεύτερης έκθεσης εποπτείας και επίσης έχουμε και τον κύριο Ροπ Ράιτ το διευθυντή της Europol, που ξαναυποδεχόμαστε στην ε, Επιτροπή μας. Θα σχολιάσει περαιτέρω τα πορίσματα αυτά της δεύτερης εποπτικής έκθεσης. Πρώτα λοιπόν θα ακούσουμε τον κύριο Ράιχαρτ Πρίμπε, το Διευθυντή Εσωτερική Ασφάλειας τη Γενική Διεύθυνσης ε, Home. Έχετε το λόγο, κύριε Πρίμπε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτές, Κυρίε και κύριοι, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις στη συμφωνία EFTP. TFTP με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ηλικία δύο ετών πλέον αυτή η συμφωνία και αρκετή εμπειρία έχουμε συλλέξει ως προς την εφαρμογή της. Θα ήθελα λοιπόν για τη Συμφωνία Οικονομικού Εντοπισμού Τρομοκρατών να σας πω ότι θα παρουσιαστούν και στα σχόλια της Europol κάποια στοιχεία με την έκθεση της αρχής τοπτείας ε, της Europol. Στο άρθρο 13 της συμφωνίας έχουμε το σύστημα των ε, ε, ενδιάμεσων εκθέσεων ε, και θα παρουσιαστεί σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η πρώτη, όπως ξέρετε, έκθεση έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο πέρυσι με την έκδοση της εκθέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάρτιο του 2011. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε για να προχωρήσουμε σε μια διεξοδική, δεύτερη διεξοδική επισκόπηση, αναθεώρηση τον Οκτώβριο εφέτος, δηλαδή λίγο μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την διαγραφή, απάλληψη όλων των δεδομένων που έχουν ηλικία ανά των δύο ετών και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία και να σας παρουσιάσουμε την έκθεση αναθεώρησης στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μέσα στο 2012 όπως είχαμε προεξαγγείλει με την πρώτη μας έκθεση. Είναι ανοιχτό το θεματολόγιο στις αναθεωρήσεις αυτές. Θα έχετε ασφαλώς και εσείς μια ευρύτερη τοποθέτηση να κάνετε. Είχαμε επικεντρωθεί στην πρώτη αλλά και στη δεύτερη αναθεώρηση τοποθετούμεθα σε θέματα που είχαν προκύψει με την υλοποίηση της ε, συμφωνίας και οπωσδήποτε θα πρέπει και με τη δεύτερη να επισέλθουμε στις πρώτες λεπτομέρειες και να εξετάσουμε τι συνέχεια, τι τύχη είχαν οι συστάσεις που είχαμε διατυπώσει με την πρώτη έκθεση. Και βέβαια σε αυτό θα ε, ενσωματωθεί και ο μηχανισμός επαλήθευσης του άρθρου 4 της Europol για να εξετάσουμε και τη λειτουργία του μηχανισμού ελέγχου. Θα προτείνουμε στην Αμερικανική πλευρά να εξεταστούν και όλα τα άρθρα της συμφωνίας που έχουν να κάνουν με αμοιβαιότητα. Θα ζητήσουμε λεπτομέρειες πληροφορίες για την υλοποίηση της συμφωνίας. Η έκθεση ασφαλώς είναι ανοιχτή όπως και αναθεώρηση σε σχόλια και συστάσεις και από τις δύο πλευρές. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω την έκβασή της. Πάντως ε, μπορούμε να πούμε ότι η συμφωνία λειτουργεί ικανοποιητικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο των Οικονομικών ε, των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν τακτική ε, και επικοδομητική επαφή έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ε, την ε, απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος οικονομικού εντοπισμού τρομοκρατών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ και στο περιθώριο αρκετών ε, ευρωαμερικανικών υπουργικών διασκέψεων έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέματα που μας απασχολούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αναθεώρηση αυτής της συμφωνίας, της εφαρμογής συμφωνίας, δεν είναι απλώ ένα γεγονός που λαμβάνει χώρα μια φορά το χρόνο ή κάθε τόσου μήνες. Είναι μια ουσιαστική ε, συζήτηση και διάλογος με τι Αμερικανικέ Αρχές με επικοδομητικό τρόπο. Θα ήθελα πολύ σύντομα να σα δώσω κάποιες ε, πληροφορίες για την εποπτεία. Λειτουργεί ικανοποιητικά το σύστημα από το Μάιο του 2001 έχει γίνει εντατική κατάρτιση των ε, εποπτών, δεν διορίζονται από την Επιτροπή. Όσοι είναι του SWIFT, οι επόπτες του SWIFT ε, συμμετέχουν και σε μέτρα κατάρτισης, σε προγράμματα κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Επίσης έχουν θεσπιστεί ε, συνθήκες για την ε, διευκόλυνση του έργου του επόπτη και του Ευρωπαίου επόπτη κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θα τα δούμε και αυτά στην αναθεώρησή μας. Για δε την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ε, οικονομικού του τρομοκρατών πρέπει να πούμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία βέβαια για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος και προσπαθούμε να ενισχύσουμε περισσότερο και να βελτιώσουμε τον μηχανισμό διασφαλιστικών δικλείδων. Είναι το έργο αυτό τεχνικού χαρακτήρα απαιτητικό και δεν μπορεί μόνο ε, με χρονικά όρια να εξεταστεί. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι μια δουλειά την οποία θα κάνει κανείς ε, σε ωράριο Εργασία τακτικό, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις άδειες και τις ασθένειες, τις απουσίες κτλ. Επίσης ε, υπάρχει και μια ομάδα εποπτών μερικής απασχόλησης, τους οποίους βεβαίως παρακολουθεί ο συντονιστής της ομάδας. Μετά τις εντατικές συνομιλίες λοιπόν το 2012, αρχές του 2012, θεσπίζεται και ένα δεύτερο, μια δεύτερη θέση στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έτσι ώστε να στηρίξει ως αναπληρωτής τον ε, επόπτη από την Αμερικανική πλευρά και αντίστοιχα χρειάστηκε και από ευρωπαϊκή πλευρά. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, δείχνουν ευαισθητοποίηση απέναντι στη σημασία τη αποτελεσματική και πρόσκοπτη λειτουργία του συστήματο των ασφαλιστικών δικλείδων. Εφέτο το Μάιο επίση ξεκίνησε μια διαδικασία για την ε, πρόσληψη του αναπληρωτή επόπτη. Δεδομένου όμως ότι είναι και πολύ λεπτό το καθήκον και σοβαρό, με απέτηση για ιδιαίτερες γνώσεις, χρειάζεται να πρόκειται για ένα άτομο το οποίο θα έχει ε, προϋπηρεσία και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τις τεχνικές γνώσεις και βέβαια απόλυτη κατανόηση και ευαισθητοποίηση επάνω στους μηχανισμούς ε, των διασφαλιστικών δικλείδων. Ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και θα αναλάβει τα καθήκοντά του, δηλαδή λίγο πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης, από την έναρξη δεύτερης ε, Το άρθρο 4 επίσης, κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, αφήνει στη Europol το καθήκον να ε, εξετάσει εάν τηρούνται τα κριτήρια από πλευρά των ΗΠΑ. Μια ειδική μονάδα της Europol έχει αναλάβει το καθήκον αυτό σε συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Θα ήθελα ωστόσο τις λοιπές λεπτομέρειες ε, να τις αφήσω για την έκθεση αναθεώρησης και για τη λειτουργία αλλά και για τη συμμετοχή της Europol. Μπορώ να τα παρουσιάσω ο κύριος Rob Wainwright εδώ μεταξύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρίμπε για την παρουσίαση που μας κάνατε. Θα ακούσουμε τώρα την Ιζαμπέλ Κρούς που θα μας παρουσιάσει τα πορίσματα της ε, κοινή ε, αρχής ελέγχου της Europol, της GSB. Παρακαλώ κυρία Κρούς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω αυτή τη δεύτερη έκθεση ε, εποπτικού ελέγχου που έγινε για το σύστημα οικονομικού εντοπισμού τρομοκρατών και τη σχετική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Παρουσιάσαμε την πρώτη έκθεση εδώ. Η έκθεση αυτή έχει γίνει τον Οκτώβριο του 2010. Μία πρώτη επιθεώρηση, ένας πρώτος έλεγχος, προκειμένου ήδη να εντοπιστούν κάποια κρίσιμα σημεία σε ό,τι αφορά το, τα δεδομένα και τα, τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 4. Επ' λοιπόν εξετάσαμε την σωστή εφαρμογή του άρθρου 4 της συμφωνίας. Και παρά τις ε, επιφυλάξεις που είχαμε στον πρώτο αυτό έλεγχο, ακριβώς εξαιτία του, του γεγονότος ότι λίγες μέρες πριν τη διενέργεια του ελέγχου ε, η Ευρωπόλ χρειάστηκε να διαβαθμίσει ως ε, από, άκρος απόρριτο το θέμα αυτό μετά από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, οπότε χρειάστηκε να κριθεί εμπιστευτική και έκθεσή μας, απόρριτη. Πάντως στο δεύτερο έλεγχο υποβάλαμε μία έκθεση με, τεσ... με πέντε θεμελιώδεις συστάσεις με τα σημεία που έχρισαν διόρθωσης κατά τη γνώμη μας για να εφαρμοστεί πλήρως το άρθρο 4 της συμφωνίας. Το Νοέμβριο του 2011 έγινε η δεύτερη αυτή επιθεώρηση, ο δεύτερος έλεγχος για να ελεγχθεί κατά πόσο είχε δοθεί μια συνέχεια στις αρχικές συστάσεις. Εξετάστηκε η εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 4 και των άρθρων 9 και 10 της συμφωνίας. Ο έλεγχος μας αφορούσε και τις ε, συγκεκριμένες ετάσεις, ε, ε, το θέμα της ασφάλειας και όλα τα συναφή με τη συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις ε, και τα κριτήρια του άρθρου 4, η κοινή Αποπτική αρχή της ε, Ευρωπόλ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τις πέντε στάσεις που υποβάλαμε, οι δύο πρώτες έχουν τηρηθεί. Σε ό,τι αφορά δηλαδή την επέμβαση του επόπτη προστασίας δεδομένων με θεσμοθετημένο και επίσημο τρόπο και συνεκτικό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης ε, είχε υλοποιηθεί και η δεύτερη μας σύσταση, ενώ οι τρεις υπόλοιπες συστάσεις που σας είχαμε παρουσιάσει πέρυσι δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ε, ενσωμάτωσή τους. Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 4 καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο επόπτης ε, ε, προσωπικών δεδομένων έχει θεσμικό πια ρόλο στην ανάλυση των αιτήσεων, οπότε η γνώμη του λαμβάνεται υπόψη και η παρουσία του εξασφαλίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Παρ' όλα αυτά, διαπιστώνουμε ότι σε σχέση με την γνωμοδότηση που είχε δώσει ο επόπτης για το πρώτο αίτημα, τα ζητήματα που επισημάνθηκαν εκεί δεν ε, διαθετήθηκαν. Κάτι που σημαίνει κατά τη γνώμη μου ότι δεν έχουν ρυθμιστεί αυτά τα θέματα. Γιατί αν είχαν λυθεί αυτές οι εκκρεμότητες, η γνωμοδότηση του επόπτη προσωπικών δεδομένων ως προς το αίτημα θα ήταν θετική. Κάτι που δεν συνέβη. Επίσης, διαπιστώνουμε μια άλλη πραγματικότητα ότι μέχρι στιγμής όλα οι αιτήσεις που υπευλήθησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες έτυχαν ε, θετικής υποδοχή από την Ευρωπόλ και έγιναν δεκτές. Ω προ την τεκμηρίωσή τους ε, θεωρούμε ότι η τεκμηρίωση αυτών των αιτήσεων δεν ήταν ε, απόλυτος επαρκής γιατί ήταν γενική Επίσης, δεν υπάρχουν περιορισμοί ε, της γεωγραφικής εμβέλειας. Οπότε καλύπτεται ο κόσμος ολόκληρος ε, στη συμφωνία αυτή για τη μεταφορά των δεδομένων, για τη μεταβίβαση των δεδομένων και για τα μηνύματα που παράγει το SWIFT. Δεν υπάρχει κανένας γεωγραφικός περιορισμός. Επίσης, ε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι αιτήσει αυτές καλύπτουν ε, όλη την περίοδο του μήνα και γίνονται ανά μήνα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Είναι μηνιαίες λοιπόν αυτές οι αιτήσει και υπάρχει μια συνέχεια σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που αποστέλλονται. Από την αρχή δηλαδή της διαδικασίας ε, υποβάλλονταν μηνιαίως αιτήσει από τον Ιούνιο του 2010 ε, μόνο τον Ιούνιο είχαμε δύο, ε, ε, το καλοκαίρι δύο. Συνήθως είχαμε κάθε μήνα το, την υποβολή αιτήματο, μάλιστα με το ευρύ γεωγραφικό πεδίο που σας περιέγραψα. Τα μηνύματα βέβαια δεν είναι τα ίδια, είναι διαφορετικά. Επίσης παρατηρήθηκε μια σχετική μείωση των μηνυμάτων, αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, ότι θέλονται περισσότερα στοιχεία, περισσότερα προσωπικά στοιχεία, μετεβάζονται λιγότερα προσωπικά στοιχεία ή όχι. Δεν είμαστε σε θέση να το κρίνουμε. Επίσης ελέγχθηκαν κάποια ε, αιτήματα μεταβίβαση στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα μηνύματα που υποβλήθηκαν για την πλήρη αποστολή δεδομένων Έχουμε ε, έχουμε ζητήσει συγκεκριμένες πληροφορίες από τι ΗΠΑ, ακριβείς και ενημερωμένε και όχι γενικές Και παρόλο που έχει διαπιστωθεί μια αύξηση των πληροφοριών που χορηγούνται από τις Ηνωμένε Πολιτείε, στην πράξη οι πληροφορίες αυτές είναι ε, ανοιχτές προς το κοινό, είναι προσιτές και πολλές φορές δεν είναι καν ενημερωμένες. Πρόκειται για παροχημένες ε, πληροφορίες, για περιστατικά που συνέβησαν πριν από πολύ καιρό και επίσης και είναι και ειδικέ πληροφορίες για κάθε συγκεκριμένη αίτηση. Είναι απλώς ένα copy-paste, μια αντιγραφή και επικόλληση απαντήσεων που είχαν δοθεί σε προηγούμενα αιτήματα. Αυτές ήταν κάποιες ε, κριτικές που ασκήσαμε στον προηγούμενο έλεγχο και από τη στιγμή που δεν ε, ε, δόθηκαν τεκμηριωμένα στοιχεία για το αίτημα, δεν ε, μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε και σωστό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή η Europol μας λέει ότι οι προφορικές αρχικά πληροφορίες περιλήφθηκαν και σε γραπτή μορφή. Οπότε έχουμε πολύ περισσότερες σελίδες με πληροφορίες που συνοδεύουν το κάθε αίτημα αλλά συνεχίζονται οι εμπιστευτικές συναντήσεις που έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στους ελέγχους που πραγματοποιεί η Europol. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα για την κοινή αποπτική αρχή της Europol, γιατί από τη στιγμή που δεν έχουμε γνώση αυτών των πληροφοριών, δεν μπορούμε να ελέγξουμε το κατά πόσο είναι περιστατωμένες. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα του άρθρου 9, τις αυθόρμητες δηλαδή πληροφορίες, δεν έχουμε ε, καταγράψει τίποτα αξιοσημείωτο. Διαπιστώσαμε ποιο είναι ο το συνολικός αριθμός των ε, ανακοινώσεων που είναι σχετικά μικρός δεδομένου, του όγκου των ε, δεδομένων που έχουν αποστείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αιτήματα του άρθρου 10, δηλαδή τα αιτήματα που γίνονται για επαλήθευση στοιχείων του συστήματο οικονομικού εντοπισμού τρομοκρατών στις ΗΠΑ. Είχαμε έξι ε, αιτήματα το πρώτο εξάμεινο και στην υπόλοιπη περίοδο επιβλήθησαν 65 επιπλέον αιτήματα. Μέχρι στιγμής δηλαδή 71 αιτήματα έχουν υποβληθεί. Είτε από κράτος μέλος, είτε από τα κράτη-μέλη, είτε από την Europol. Μιλούμε για τεράστιο όγκο πληροφοριών. Μπορεί ο αριθμός των ετοιμάτων να είναι ε, μεγάλος, αλλά από άποψη προστασίας δεδομένων δεν έχουμε να επισημάνουμε τίποτα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι η Europol έστειλε μια επιστολή στην Κοινή Εποπτική Αρχή, την GSP, δεδομένου ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών είχε ζητήσει πρόσβαση στην έκθεσή μας και αυτό εξετάστηκε στην τελευταία ολομέλεια τελικά η κοινή εποπτική αρχή ε, δεν ε, αντιτάχθηκε στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δημοσίευση, για χορήγηση της έκθεσής μας στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Κατά τη γνώμη, στο, κατά μας, ε, στην έκθεση εκείνη δεν υπήρχε τίποτα, καμία επιχειρησιακή πληροφορία που θα μπορούσε να αντιβαίνει στην ανάγκη να δημοσιευθεί η έκθεση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ας ακούσουμε τώρα τον διευθυντή της Europol, τον κύριο Ρόμπ Wainwright. Παρακαλώ κύριε Wainwright. Γεια σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω το λόγο πάνω σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ επίσης και την GSP και την Επιτροπή, όχι μόνο για αυτά που είπαν σήμερα, αλλά και για τις συνεχιζόμενες συστάσεις και σύμβουλες που αφορούν κάποια τμήματα της συμφωνίας αυτής. Με το JSP τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε συνεργαστεί στενότατα και έπαιξαν σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση της κατάστασης. Ο μόνος επίσημος μηχανισμός προβλέπεται στα πλαίσια του άρθρου 13 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εμπειρία μας εδώ μας λέγει ότι η αναθεώρηση αυτό που συζητάμε σήμερα δεν είναι κάτι που θα πρέπει να αντικαταστήσει το 2013. Πέρυσι μου ζητήσατε να σχολιάσω την πρώτη έκθεση του JSP. Σας έδεσα αρκετά λεπτομερείς πληροφορίες για το ρόλο της Europol στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής Επαναλαμβάνω φέτος ότι οι πληροφορίες που πήραμε πέρυσι ισχύουν και σήμερα, καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων στους τομείς αυτούς και διορθώνουν και ορισμένες παρανοήσεις οι οποίες είχαν έρθει στην επιφάνεια σχετικά με τον τρόπο λειτουργία της συμφωνίας. Την προηγούμενη εβδομάδα έστειλα μια επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής για να σας ενημερώσω καλύτερα για το πώς εργαζόμαστε και να σας ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουν λοιπόν καταστεί διαθέσιμες πάρα πολλές πληροφορίες προς την Επιτροπή σας άνω του επίπεδου απλής περιγραφής των, της λειτουργίας, κάτι το οποίο έρχεται ε, σε σχέση φυσικά ε, με την προστασία του κοινού συμφέροντος και την ε, διαφανή λειτουργία της Αεροπόλου. Κανείς δεν αρνείται ότι υπάρχουν ευαισθησίες στα πλαίσια της λειτουργίας αυτής της συμφωνίας, όπως επίσης και το θέμα των ευαίσθητων πληροφοριών και εκεί ακόμα θέλουμε να λειτουργούμε με διαφανή τρόπο. Ασχολούμεθα κυρίως με το αίτημα δημόσιας πρόσβασης, το οποίο εστάλει στην Ευρωπόλ εδώ και λίγες εβδομάδες για την πρόσβαση στην πλήρη απόρριτη μορφή της έκθεσης αυτής. Όπως είπε ο κ. στην επιστολή του, το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Έχουμε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο το οποίο θα έλεγα δέχεται την αρχή της δημόσιας πρόσβασης μαζί με την αρχή της προστασίας των δεδομένων που θα βλάψουν την λειτουργία της Ευρωπολ και των εταίρων της. Το αίτημα το οποίο έχουμε στα πλαίσια της λειτουργίας μας να διαβουλευόμεθα με τρίτα πλευρές, ε, των οποίων οι εργασίες ε, θα φύγονται από την δημοσιοποίηση Κυρία Κρούζ, εδώ δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Εμείς ήρθαμε σε επαφή και με τις Ηνωμένε Πολιτείες γιατί από εκεί προέρχονται τα περισσότερα από τα ευαίσθητα στοιχεία στα οποία αναφερόμαστε στην έκθεση. Περιμένουμε την τελευταία γνωμοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Την προηγούμενη εβδομάδα συζήτησαν σε ολομέλεια τα θέματα αυτά και μας επέτρεψαν ήδη να μοιραστούμε την έκθεση JSP με τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, γιατί δεν είχαν διαβάσει την έκθεση αυτή. που να το κάνουν δεν θα έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν αιτήσει για δημοσιοποίηση. Εδώ και λίγες μέρες λοιπόν ε, πήραν την έκθεση αυτή και θα μας ε, την σχολιάσουν το ταχύτερο δυνατόν και έτσι τότε θα μπορέσω να ικανοποιήσω το αίτημα του κυρίου Λόπες Αγγουιλάρ. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ενημερώσω την, λειτουργία, την Επιτροπή για τη Λειτουργία της υπηρεσίας μας σχετικά με τις παρατηρήσεις κυρία Σκρούς. Όπως γνωρίζετε η συμφωνία αυτή σχετικά με την Ευρωπόλ έχει τρία άρθρα. Καταρχάς επαλήθευση λειτουργίας και το άρθρο έχει σημασία να πω ότι εμείς δεν βλέπουμε τα δεδομένα τα οποία μεταφέρονται από ένα συγκεκριμένο παροχέα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είμαστε φυσικά υπεύθυνοι για τις άλλες ρήτρε ασφαλείας που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία για τις πιθανές έρευνες και παρεμβάσεις στη μεταφορά των δεδομένων. Αυτά είναι εξίσου σημαντικά με ό,τι αναφέρεται στο άρθρο 4 και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν ένα συνολικό πακέτο. Έχω την αίσθηση ότι δημιουργείται συχνά μία παρανόηση. Όταν αδειοδοτήσουμε τη μεταφορά δεδομένων στα πλαίσια του άρθρου 4, το σύνολο των δεδομένων αυτών είναι διαθέσιμα στις Αμερικανικές αρχές. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι τρόποι εφαρμογής των υπολείπων ρητρών ασφαλείας. Μόνο ένα πολύ μικρό τμήμα των δεδομένων αυτών ε, παρέχεται προς πρόσβαση στους Αμερικανούς. Σχετικά με το άρθρο 9 τώρα. Αυτό επιτρέπει στις Ηνωμένε Πολιτείε να δίδουν προς την Europol αυθόρμητα τα αποτελέσματα των ερευνών τους και τη δυνατότητα ε, εμείς να ζητούμε τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν, από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία εδώ και δύο χρόνια, υπήρξαν 24 αιτήματα επί τη βάση του άρθρου 4 από πλευρά. ήπα Σε έξι τέτοιες περιπτώσεις δεν δεχθήκαμε εμείς το αρχικό αίτημα, εκτός και αν αποκτήσουμε από πλευρά των Αμερικανών επιπλέον τεκμηριώσεων και δικαιολογιών. Για το άρθρο 9, αυθόρμητη ενημέρωση, έχει οδηγήσει από πλευράς Αμερικανών σε 54 περιπτώσεις σε έρευνες που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη η Ευρωπόλ ζήτησε από πλευρά Αμερι... τους... τους Αμερικανούς 93 φορές να προχωρήσουν σε έρευνες που οδήγησε σε 300 ε, περίπου συνδέσμους ε, ενημέρωσης σχετικά με τα τρομερά γεγονότα στην Νορβηγία το 2011 τον Ιούλιο με μεγάλη απώλεια ζωής. Άμεσα εμείς υποβάλαμε τρία αιτήματα άρθρο 10 στις Αμερικανικές υπηρεσίες για να υποστηρίξουν τις τρέχουσες διαδικασίες έρευνας στην Ευρώπη. Ταχύτατες απαντήσεις από πλευρά των Αμερικανών οδήγησαν την Ευρωπόλ να εντοπίσει άτομα, πηγές χρηματοδότησης και υποστηρικτές του Μπράιβικ. Χρησιμοποίησαμε τα στοιχεία αυτά λοιπόν και να αποκαλύψουμε ένα περίπλοκο και ευρύτατο δίκτυο χρηματοδότησης διεθνές. Οι πληροφορίες επίσης ήταν πολύ σημαντικές και για τη λειτουργία του δικτύου πρώτης απόκρισης ε, της Europol που εφαρμόστηκε, τέθηκε σε λειτουργία στην Νορβηγία. Οδηγηθήκαμε στην ανακάλυψη πολλών ε, λογαριασμών τραπεζικών άμεσα στο όνομα του υπόπτου ή και στο όνομα εταιριών που ανήκαν στον υπόπτο. Δεδομένα επίσης ε, σχετικά με την αγορά χημικών και εξοπλισμών που αγοράστηκαν από τον Πράιβεκ στην προετοιμασία των εκρηκτικών που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Τέλος, τα δεδομένα δείχνουν ότι η λειτουργική φάση των δραστηριοτήτων του υπόπτου μπόρεσε να διαφωτιστεί από τους μηχανισμούς τους οικονομικούς που χρησιμοποίησε για να προπαρασκευάσει τις επιθέσεις του. Χωρίς το μέσο αυτό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε. Ήταν σημαντικό λοιπόν, ιδιαίτερα λόγω του κατεπήγοντος χαρακτήρα της έρευνας, και γιατί θελήσαμε άμεσα να δούμε αν ο Μπράιβεκ λειτουργήσε μόνος του ή ήταν τμήμα μιας παγκόσμιας ακροδεξιάς συνωμοσίας. Στρέφομαι τώρα στις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο χρόνο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Πρώτον θα ήθελα να πω ότι η από κοινού αντιμετώπιση της Επιτροπής και της JSP επηρέασαν αρνητικά την βελτίωση της διαδικασίας επί τη βάση του άρθρου 4. Ο τρόπος με τον οποίο μπορέσαμε να αμφισβητήσουμε τους Αμερικανούς έτσι ώστε να μας δώσουν όλες τις απαιτούμενες τεκμηριώσεις και εξηγήσει, ιδιαίτερα τον πρώτο χρόνο, οδήγησε σε περαιτέρω εκλεπτισμένες πηγές πληροφορίας που βελτίωσαν την ποιότητα των Αμερικανικών ετοιμάτων και θα ήθελα να πω ότι είχαμε πάρα πολύ θετική ανταπόκριση από πλευρά των Αμερικανικών αρχών στα πλαίσια της εφαρμογής της συμφωνίας. Υπήρξε πρόοδος, αυτό αναγνωρίστηκε από το JSP, την αρχή εποπτείας. Και αυτό δείχνει τις τεράστιες προσπάθειες οι οποίες έγιναν από την Ευρωπόλ τα τελευταία χρόνια για τα συγκεκριμένα προβλήματα. Συνεργαστήκαμε όχι μόνο με το JSP αλλά και με τους αρμόδιους ε, υπαλλήλους και υπευθύνους μάλλον για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Κάναμε ομάδες εργασίας για να ελέγξουμε τον τρόπο λειτουργίας της συμφωνίας και εποφεληθήκαμε με οδήποτε τρόπο μπορέσαμε από τις συνθήκες για να βελτιώσουμε τη συμφωνία αυτή σε εφαρμοστικό επίπεδο μετά από την αξιολόγηση της πρώτης έκθεσης του JSP και μετά από συζητήσεις που έγιναν εδώ, λεπτομερέστατες συζητήσεις στα πλαίσια πνεύματος συνυπευθυνότητας επικοδομητικής και υπεύθυνη ανάμεσα σε ισότιμους εταίρους. Σχετικά με τη δεύτερη έκθεση JSP, η Αεροπόλ επίσης ε, έκανε σχόλια στην πρώτη έκθεση. Κάποιες από αυτές δεν αντικατοπτρίζονται στην τελική έκθεση και αναφέρομαι σε αυτές σήμερα, όπως είπε η κυρία Κρούς μετά από τις πέντε αρχικές συστάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην έκθεση, δύο έχουν εφαρμοστεί πλήρως, η τρίτη έχει αν πολλής, ε, αν θέλετε, εφαρμοστεί κατά τη γνώμη μας, αλλά αναμένεται να ελεγχθεί τεχνικά από το JSP και δύο βρίσκονται σε φάση εφαρμογής. Στην επίσημη δήλωση το JSP αναφέρθηκε στο ρόλο του υπεύθυνου για τα προσωπικά δεδομένα. Θέλω να πω ότι ο συγκεκριμένος ε, αρμόδιος ε, είναι σε επαφή μαζί μας, στενή επαφή, ανταποκρίνεται σε όλα μας τα αιτήματα μια νέα μορφή των λειτουργικών οδηγιών στα πλαίσια της λειτουργίας του JSP για την ενίσχυση του τρόπου λειτουργία μας ε, συνεχίζει να εφαρμόζεται. Να τονίσω εδώ ότι οι θετικές αποφάσεις σχετικά με το 4, το άρθρο 4 δεν ελήφθησαν μετά από αντίθετη άποψη του DPO. Αντίθετα πήραμε μέτρα για να διευκρινιστεί το DPO και ο συγκεκριμένος υπεύθυνο λοιπόν προσωπικών δεδομένων μας είπε ότι παρακολουθεί από κοντά την εφαρμογή του JSP και την εφαρμογή μάλλον των συστάσεων του JSP και είναι ικανοποιημένος κατά τη γνώμη του όλες οι συστάσεις της JSP εφαρμόστηκαν όσο καλύτερα μπορούσε η Αεροπολ στα πλαίσια και της εξάρτησης αλλά και συνεργασίας ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Κύριε Γουένραϊτ, έχουμε ένα θέμα χρόνου. Έχουμε ένα χρονικό πλαίσιο και ένα χρονικό περιορισμό, παρακαλώ μην το αγνοήσετε αυτό. Αυτό το σημείο ε, δεν πρέπει να ξεπεράσει ένα χρόνο, αλλά θα ήθελα να ζητήσω την υπομονή και τη γενεοδορία των διερμηνέων επανειλημμένα. Αλλά δεν θέλω να γίνεται συστηματικά αυτά. Γι' αυτό παρακαλώ να παρουσιάσετε την υπόλοιπη ομιλία σας με συνθετικό τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε και χρόνο ομιλίας που είναι και το ζητούμενο. Σα ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και για τη δική μου την οργάνωση και θέλω να βεβαιωθώ ότι έχει στη διάθεσή της κάθε λεπτομέρεια η Επιτροπή, αν μου επιτρέπετε, θα συνοψίσω. Για κάποια άλλα σχόλια, τα οποία υπεγράμμισε και ο Πρόεδρος, ε, το άρθρο 4 ορίζει ένα χρονικό πλαίσιο και θα ήθελα σε αυτό να αναφερθώ στη φύση της τρομοκρατικής που ε, αφορά τις, ε, που εξετάζουν οι έρευνές μας, το χρόνο της, ε, του προγραμματισμού δηλαδή. Και δεν μπορούν να αποκλειστούν τέτοιες δραστηριότητες προληπτικές από την περίπτωση της προετοιμασίας. Όσον αφορά τη χρήση προφορικών πληροφοριών. Δεν ισχύει ο ισχυρισμό ότι στηριζόμαστε σε μη και καταδιαγραμμένε προφορικές ε, δηλώσεις ε, για, ε, για τα αιτήματά μας, δυνάμει το άρθρο 4. Είχαμε τέσσερι συνεδριάσει με την Αμερικανική πλευρά. Εμείς στηριζόμαστε σε γενικές ενημερώσεις, briefing δηλαδή με την Αμερικανική πλευρά, με παρουσία όλων των εμπλεκομένων εταίρων, ώστε να γνωρίζουμε όσο δυνατόν καλύτερα το... και να γνωρίζουν όλη τη βάση πάνω στην οποία λαμβάνονται οι αποφάσει μα. Για να ολοκληρώσω, είμαι πεπισμένο ότι η Europol έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να έχουμε όλα τα στοιχεία για να λαμβάνουμε αποφάσει και συμφωνίε. Έχουμε φτάσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο μέχρι τώρα τουλάχιστον υλοποίηση. βελτίωση χωρί ασφαλώ, αλλά δεν ξέρω πόσοι γιατί είναι πάρα πολύ εντατική η δουλειά που κάνουμε με τέσσερα workshops ε, τακτικά με την GSP και, τους, ε, την Αμερικανική πλευρά. Στο πλαίσιο που μας ε, επιτρέπει τουλάχιστον νομοθεσία και στην πλαισίωση αυτή νομοθετική, δεν ξέρω αν μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητά μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε φυσικά και προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας της καταπολέμησης τρομοκρατίας. Παρακαλώ. Κυρίε και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για ερωτήσει. Η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα περιοριστώ και εγώ σε δύο σημεία. Ένα το οποίο και η κυρία Κρούς ανέφερε ως προς τα αιτήματα της αμερικανικής πλευράς, όπου είναι ανεπαρκής η αιτιολόγηση και ασαφές το αίτημα. Δεν θέλω να κάνω υποθέσεις για το πού οφείλεται αυτή η ασάφεια ή Φερρυπίν γιατί δεν έχουν ε, ε, συγκεκριμένα στοιχεία ή γιατί δεν θέλουν να διατυπώσουν πιο συγκεκριμένα αιτήματα οι Αμερικανοί έτσι ώστε να έχουν πιο ευρεία αποστολή δεδομένων από πλευράς μας. Και πάντως θα ήθελα να επισημάνω ότι πρόκειται και για μη πρακτικό τρόπο αλλά και για παραβίαση της συμφωνίας καθαρά γιατί ορίζει ότι θα πρέπει ως το δυνατόν πιο συγκεκριμένα και με στενό ε, πεδίο να διατυπώνονται τα αιτήματα των Αμερικανών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό το στόχο. Θα ήθελα στόσο και να σας ε, συγχαρώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ηνωμένες Πολιτείες διότι χρειάστηκαν μόνο δύο χρόνια έτσι ώστε να συμφωνήσουν σε αυτό το οποίο έλεγα εγώ εξ αρχής ότι χρειάζεται μόνο ένα επόπτης, ένα αρμόδιος για τον έλεγχο από τις δύο πλευρές. Σας ε, συγχαίρω λοιπόν, τα καταφέρατε εν τέλει. Κύριε Φως. Ευχαριστώ. Από ό,τι ακούω, από τις ε, παρουσιάσεις σας. Υπάρχουν βελτιώσεις, υπάρχουν κάποιες αλλαγές ε, βάσει των προτάσεων του JSP από το πρώτο κομμάτι, αλλά και περαιτέρω βελτιώσεις χρειάζεται ασφαλώς να πραγματοποιηθούν. Χαίρομαι που έχουν αναλάβει καθήκοντα οι DPOs και θα προχωρήσουν φαντάζομαι με τις σχετικές διαδικασίες. Έχω την αίσθηση ότι χάρη και στη δική μας τη συμφωνία για το πρόγραμμα αυτό, για το σύστημα οικονομικού εντοπισμού τρομοκρατών, μπορούμε να έχουμε πιο συγκεκριμένα δεδομένα, γιατί προσπαθούν και οι δύο πλευρές από ό,τι φαίνεται να τηρήσουν ως το δυνατόν πιο πιστά και αυστηρά τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί με τη συμφωνία. Και μια μικρή συμβολή μάλλον από πλευρά μου, όταν επισκεφθήκαμε το Υπουργείο των οικονομικών και για την περίπτωση και για, για, την επίθεση, για τις επιθέσεις στην Τουλούζη, ε, είδα πολύ συγκεκριμένα αυτές οι αναλύσεις τι μπορούν να προσφέρουν και σε γνώσεις και σε πρόοδο για, ε, για την ανάκριση για την διερεύνηση μιας υπόθεσης. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να έχουμε πολύ καλή προόδο ακόμη και σε ευαίσθητα θέματα και σε διαβίβαση για ευαίσθητες υποθέσεις και περιπτώσεις προσωπικών δεδομένων. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι είδου προσδοκίες μπορείτε να έχετε ως προς την ικανοποιητική ή επαρκή πάντως προστασία δεδομένων έτσι ώστε ταυτόχρονα εξυπηρετείται και ο στόχος της ασφάλειας μια, εξο... μια αξιολόγηση την οποία από την κυρία Κρούς περιμένω μάλλον να ακούσω γιατί ξέρουμε ότι έχει προχωρήσει καλά η Europol έχει κάνει σημαντικές βελτιώσεις όπως διατυπώνεται όπως διαπιστώνεται ε, αλλά χρειάζονται βέβαια και κάποιες άλλες μέχρι ό,τι μπορούμε να πούμε σταθμίζοντας την κατάσταση ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι Φυσικά πρέπει να δούμε και τι είδου προσδοκίε μπορεί να έχει κανεί για το μέλλον. Φέρει περισσότερη διαφάνεια αλλά πάντως νομίζω ότι μπορούμε να πούμε εν γέννη ότι επικρατεί αίσθηση ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά καλά. Έχει αρχίσει το σύστημα να λειτουργεί ικανοποιητικά και για την ανταλλαγή των δεδομένων και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η κυρία Νετφέλτ. Πρόεδρε, έχω και εγώ κάποιες ε, παρατηρήσεις. Τώρα συγγνώμη για την βραχνή μου φωνή. Δύο παρατηρήσεις καταρχάς για τη διαδικασία Είμαι εδώ σήμερα ως μέλος του Κοινοβουλίου για να κάνω τη δουλειά μου, δηλαδή να ε, ελέγξω πώς λειτουργούν οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαι εδώ για να κάτσω επί 45 λεπτά να ακούω τον κύριο Wainwright και άλλους να κάνουν παρουσιάσεις και να μην έχω χρόνο για ερωτήσεις. Και σας παρακαλώ στο μέλλον έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για να κάνουμε αυτό που είναι η δουλειά μας. Δηλαδή να κάνουμε ερωτήσεις και να ρωτήσουμε τον κύριο Wainwright και τους άλλους ερωτήσεις, οι οποίες θα λάβουμε και απαντήσεις. Πρώτον. Δεύτερον, και ερωτώ, επί τίνη βάση μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο αυτό που οφείλουμε να κάνουμε ως βουλευτές εάν δεν έχουμε την έκθεση. Και αν μας λέτε ότι έχετε αντιρρήσει και δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσει ω προ τη δημοσιοποίηση των εκθέσεων. Επομένω, ρωτώ και ω ιδιώτη, δώστε μου την έκθεση και αν χρειαστεί θα καταφύγω και στα δικαστήρια ακόμη. Θα προσφύγω και στα δικαστήρια. Μου φαίνεται απαράδεκτο να δίνουμε στοιχεία μαζικά σε ξένες χώρες, αλλά να μην ενημερώνουμε τους πολίτες και τους βουλευτές, ε, κύριε Γουέινραιτ, για τα δεδομένα αυτά και το πώς χρησιμοποιούνται από άλλους. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να ζητώ την άδεια των Ηνωμένων εγώ ή εμείς για να εφαρμόσουμε τις δικές μας προδιαγραφές διαφάνειας, γιατί αν θα πάντοτε από μια τρίτη χώρα για το κατά πόσον μπορούμε να δημοσιεύουμε στοιχεία, τότε ας πάμε σπίτια μας όλοι, δεν χρειάζεται να υπάρχουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Και βλέπετε ότι είμαι αρκετά ενοχλημένη από αυτήν την κατάσταση. Κύριε Wainwright, αναφερθήκατε σε πολλές λεπτομέρειες της εκθέσεως. Ένα συμπέρασμα όμως προκύπτει. Σημαντικό για τη δουλειά μας. Είναι εκεί που λέγεται ότι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η συμφωνία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν όλε οι διασφαλιστικές δικλείδε του άρθρου 4 όπω ορίζεται. Δηλαδή, παρότι έχει προσδιοριστεί αυτό το άρθρο το οποίο σε στόχο έχει να περιορίζει τα δεδομένα τα προσωπικά που θα διαβιβάζονται, διαβιβάζονται τα πάντα. Άρα τι το θέλουμε. Τι θέλουμε το άρθρο και τι θέλουμε και τι συμφωνίε. Την περάσουμε από τη μηχανή κοπή εγγράφων και τελειώνουμε. Να του δίνουμε και τα δεδομένα όσα θέλουν και τελειώνουμε. Δεν τη χρειαζόμαστε τη συμφωνία. Επίση, Κάτι ακόμη, παρατήρηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον. Εγώ υπερψήφισα, αλλά με μεγάλη δυστημία, την έκθεση αυτή με πολλούς δισταγμούς και μόνο για ένα λόγο, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είχε υποσχεθεί ότι μέσα σε ένα χρόνο θα είχαμε σύστημα εξαγωγής δεδομένων μέσα στην Ευρώπη. Πού το λοιπόν, κύριε Πρίμπε, πού είναι το σύστημα. Αυτό που προτείνατε πολύ εκ των υστέρων ήταν ένα ευρωπαϊκό σύστημα ε, οικονομικού εντοπισμού που ξεπερνά πολύ περισσότερο, κατά πολύ περισσότερο αυτό που ζητούσαν οι Αμερικανοί. Άρα έχετε προδώσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις υποσχέσεις τη Και άλλη μια τελευταία παρατήρηση, λεπτομέρεια ίσως, ότι έτυχε να μελετήσω μια ε, διατριβή επιστημονικού χαρακτήρα όπου και αν θέλετε σου και τα στοιχεία της, ε, εξετάζονται οι μέθοδοι, συγκεκριμένες μέθοδοι για τη συλλογή των στοιχείων υπό τη συμφωνία αυτή. Στο 5.3 της συμφωνίας αναφέρεται ότι θα υπάρχει data mining, δεν θα συλλέγονται δηλαδή ανεξέλεγκτα στοιχεία. Εμείς χωρίς να είμαστε ειδικοί στο ίντερνετ χρησιμοποιούμε το ίντερνετ. Θα ήθελα λοιπόν, όπως ο κάθε χρήστης, να είμαι βεβαία ότι δεν θα συλλέγονται ανεξέλεγκτα στοιχεία. Φαίνεται όμως ότι η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι ακόμη πιο... Ε, παρεμβατική, απλώ δεν έχει το, δεν έχει το όνομα data mining. Μα λέτε ότι δεν γίνεται data mining, αλλά γίνεται κάτι ισοδύναμο και χειρότερο ακόμα που δεν καταγράφεται συμφωνία και που τελικά σημαίνει ότι ακυρώνονται στην πράξη όλε ή πολλέ από τις ρήτρε για τη ασφαλιστική δίκλυδα. Ναι, μα λέτε ότι κάνετε ανάλυση κοινωνικών δικτύων κτλ. Δεν χρειάζεται να σα δώσω τώρα όλε τι σελίδες και τι λεπτομέρειε τεχνικέ, αλλά πάντω καταλήγω ότι την πατήσαμε. Μα τη στήσατε και την πατήσαμε. Δηλαδή, υπογράψαμε και δεχθήκαμε ένα σύστημα άχρηστο στην πράξη, με ρήτρε οι οποίε δεν μα είχαν γνωστοποιηθεί επαρκώ, που δεν λειτουργούν σωστά και τώρα ούτε καν μα δίνετε την έκθεση για το πώ λειτουργεί το σύστημα. I feel... Και ε, φοβούμαι ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό εδώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ε, υπογραμμίσω αυτά που είπε η Σοφία Ιντβέλτ. Δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο προσεκτικές τα λόγια τους σε άλλες ομάδες. Γιατί ρίχνοντας μια ματιά σε αυτό που έχω μπροστά μου, τη δημόσια δήλωση, όχι την έκθεση, αυτό που μας διάβασε δηλαδή η Σόφη, ότι δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες του άρθρου 4. Μα εμείς αυτό ζητήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό ψηφίσαμε όταν εξετάστηκε η συμφωνία και όταν είχαμε καταψηφίσει στην αρχική εκδοχή. Και αυτό είναι πραγματικά εκνευριστικό. Και διαβάζω παρακάτω. Αναφέρεται ότι η Europol δεν βλέπει ή διαχειρίζεται τα στοιχεία SWIFT ή το γνωρίζει το πραγματικό του όγκο. Λαμβάνει κάθε μήνα κατά μέσο όρο μία αίτηση που καλύπτει συνήθως ε, την περίοδο ενός μηνός η αίτηση αυτή. Κάτι που σημαίνει ότι οι συνέπειε της συμφωνίας, όπως λέει το κείμενο, όπως εφαρμόζεται τουλάχιστον τώρα, είναι ότι τα στοιχεία για συγκεκριμένες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ε, χορηγούνται για ένα χρονικό ε, όριο για κάθε συγκεκριμένη μέρα. Δηλαδή, εμείς ζητήσαμε ακριβώς να περιοριστεί ο αριθμός των μεταβαζόμενων στοιχείων. Και τι βλέπουμε τελικά, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο αριθμός των στοιχείων μεταβιβάζεται, το σύνολο των στοιχείων χωρίς κανένα περιορισμό όπως είπε και η Σοφή. Σίγουρα η... δεν είναι αυτή η συμφωνία που ζητούσαμε εμείς, ούτε αυτή που θέλαμε. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να έχουμε μια ευκαιρία να πούμε κάτι γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δημιουργήθηκε μια σύγχυση στη συζήτηση και τώρα λέμε, εντάξει, βρισκόμαστε πρωτοτελεσμένο γεγονότο, συγγνώμη, τελειώσαμε. Εμείς θέλουμε περιορισμό των ε, μεταβιβάσιμων στοιχείων για να είναι ε, χρήσιμη η συμφωνία, έστω και σε μία περίπτωση, πολύ αμφιβάλλω ότι είναι απαραίτητη από την άποψη της αναλογικότητας ό,τι αφορά την αξιολόγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γιατί χρήσιμο εργαλείο, όπως αναφέρει η έκθεση, δεν δικαιολογεί μια τέτοια τεράστια μαζική εισβολή στην ιδιωτική σφαίρα όλων των Ευρωπαίων πολιτών, Νομίζω ότι είναι παρατραβηγμένη η κατάσταση, σίγουρα δεν είναι αυτό που ζητήσαμε εμείς και όλα τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλες οι εγγυήσεις που ζητήσαμε στην ψηφοφορία για τη συμφωνία αυτή, φαίνεται ότι δεν έχουν τηρηθεί μετά από δύο χρόνια και βλέπετε τις συνέπειες. Δεν θέλαμε να εφαρμοστεί στην πράξη. Γι' αυτό ζητήσαμε ασφαλιστικές δικλείδες, όχι όμως κενές περιεχομένου, γιατί ζητήσαμε για κάποιο λόγο αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες, για να μην εφαρμοστεί όσοι έχει συμφωνία. Τελικά δεν εφαρμόζονται οι ασφαλιστικές δικλείδες. Το σύστημα αυτό δεν ευθυγραμμίζεται με το ε, θεμελιώδες κοινοτικό δίκαιο. Το γνωρίζουμε αυτό και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να το ελέγξουμε και να διασφαλίσουμε ευθυγράμμιση της συμφωνίας αυτής με το συνταγματικό κοινοτικό δίκαιο. γιατί αλλιώς θα χρειαστεί να προσφύγουμε κατά τη συμφωνία στο δικαστήριο. Ευχαριστώ. Η κυρία Ματιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική. Θα πω ότι είμαι ικανοποιημένη από τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας από την Ευρωπόλ. Υιοθετήθηκε από 480 ψήφους στο Κοινοβούλιο η συμφωνία αυτή μια μεγάλη πλειοψηφία κοινοβουλευτικών και δώσαμε την εφαρμογή της συμφωνίας στην Ευρωπόλ που έχει πολλές αποστολές να φέρει πέρας. Η συμφωνία αυτή λοιπόν από το 2010 εφαρμόζεται με μια αρχή ελέγχου η οποία επαληθεύει τη λειτουργία. Είναι καλό που οι Αμερικανοί και αυτοί ε, θα προσλάβουν κάποιους για να ελέγχουν και από τη δική τους πλευρά. Είμαι αρκετά ικανοποιημένη. Η αρχή ελέγχου αναφέρεται σε πέντε συστάσεις στα πλαίσια του δεύτερου ελέγχου. Από αυτές έχουν μείνει δύο ή τρεις. Δύο οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, μία η οποία εφαρμόζεται και δύο οι οποίες είναι στο πρώτο στάδιο εφαρμογής. Νομίζω ότι μετά από δύο χρόνια δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την Ευρωπόλ και ε, σίγουρα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την Ευρωπόλ για την έκθεση την οποία ψηφίσαμε εμείς. Δεν μπορεί να φταίει ο Wainwright για τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Σας θυμίζω επίσης ότι η ελεγκτική αρχή, η αρχή εποπτείας, έκανε ε, τους ελέγχους της και επίσης και ο υπεύθυνο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και όλοι είναι ικανοποιημένοι. Ας αφήσουμε λοιπόν την Ευρωπόλη να συνεχίσει στο σωστό δρόμο και θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Άκουσα πολλά για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Άκουσα πολλά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν άκουσα να μιλάμε για την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτό που με απασχολεί εμένα είναι η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Κύριε Φως, βλέπω ότι θέλεις ακόμη ένα λεπτό, μόνο ένα λεπτάκι, έτσι δεν είναι. Ναι, να προσπαθήσω, Πρόεδρε. Απλώ θα ήθελα να απαντήσω στην ε, Σοφία για την έκθεση πολύ σύντομα. Βεβαίω δεν μπορώ εγώ να κρίνω εάν μπορεί να δημοσιοποιηθεί η έκθεση ή όχι. Αλλά η κατάσταση έχει να κάνει με την ασφάλεια. Και στα εθνικά κοινοβούλια ακόμη δεν λαμβάνουμε όλα τα έγγραφα, ε, γιατί χαρακτηρίζονται ω απόρριτα, εμπιστευτικά κτλ. και μόνο εν μέρη έχει κανεί πρόσβαση. Ε, νομίζω ότι εδώ ίσως ε, να δίνεται κάπου η δυνατότητα κανείς να πάρει το έγγραφο, να πάει σε μια γωνιά να το διαβάσει διακριτικά. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν αυτά πράγματα είναι εν γέννη απόρριτα και ότι θέλουμε να δημοσιοποιούνται τα πάντα δεδομένου ότι υπάρχουν και πολλές διαρροές. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, πρέπει να δείξουμε μια κάποια κατανόηση για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι άλλοι να χειριστούν τα πράγματα. Φυσικά δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά όπως είπα και στα Εθνικά Κοινοβούλια έτσι είναι η κατάσταση. Ας αποφύγουμε συζήτηση μεταξύ μας τώρα. Ο κύριος Πρίμπε έχει το τρένο του σε λίγο. Είπε ότι οπωσδήποτε πρέπει να φύγει. Παρακαλώ και εσύ Σοφή στη δευτερολογία σου να είσαι πολύ λακωνική. Προς τον κύριο Βόσα ήθελα να πω ότι ακόμη και σε εθνικό επίπεδο δεν μπορεί οτιδήποτε τυχαία να διαβαθμίζεται ως απόρριτο. Θα πρέπει να αιτιολογείται αυτός ο χαρακτηρισμός. Ακόμη και οι ίδιοι συντάκτες της έκθεσης δεν έχουν αντίρρηση με τη μεταβίβασή της. Δεν είναι ε, κάποιες λεπτομέρειες λειτουργικές. Εμείς δεν ζητούσαμε ε, αναφορά των λειτουργικών λεπτομέρειών. Ζητήσαμε την έκθεση για την εφαρμογή μιας συμφωνίας που οι περισσότεροι απρόθυμα, με βαριά καρδιά την υπερψηφίσαμε. Και δεν μπορώ με μια τρισέλιδη σύνοψη να κάνω επαρκή έλεγχο της συμφωνίας αυτής. να υπε... Μου ζητήθηκε να υπερψηφίσω αυτή τη συμφωνία. Πώς τώρα μπορούν να μου ζητάνε να ψηφίσω για διεθνεί συμφωνίες αν ως Ευρωβουλευτής μετά δεν έχω το δικαίωμα να ελέγξω τέτοια συμφωνία. Και από τα συμπεράσματα τη σύνοψη τη τρισέλιδη, ε, έχω θορυβηθεί ακόμη περισσότερο. Αναφέρονται στα συμπεράσματα ότι είναι ουσιαστικά περίτη και άχρηστη συμφωνία, γιατί ούτω ή άλλω όλα τα στοιχεία μεταφέρονται, όλα τα δεδομένα μεταβιβάζονται. Εσεί ε, θα έπρεπε ω Ευρωβουλευτή να είχατε ανησυχήσει και να θορυβηθεί. Φυσικά και μα ενδιαφέρει η ασφάλεια. Όλοι ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια. Αλλά μια κακή συμφωνία που εφαρμόζεται και ελαττωματικά δεν εξασφαλίζει ασφάλεια. Θέλουμε μια καλή συμφωνία και σωστή εφαρμογή τη. Αυτό που αναφέρεται στα συμπεράσματα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα περιορισμό στη μεταφορά των δεδομένων. Και όλοι αναφέρθηκαν στην Τουλούζη. Ο νεαρός δολοφόνος ήδη υπήρχε στη... ήταν συσυμβασμένο στις μυστικές υπηρεσίες και παρόλα αυτά ε, είχε διαπράξει τέσσερις δολοφονίες πριν το τελευταίο μακελιό. Κοίτα και στο κατάλογο και των Αμερικανών. Γιατί λοιπόν ε, συστηματικά μας ζητάτε να συνενέσουμε στη μαζική συλλογή προσωπικών δεδομένων χωρίς ε, σε, αντιστα... αντιστάθμισμα να μας εξασφαλίζεται προστασία και ασφάλεια. Ας ακούσουμε απαντήσεις και αντιδράσεις. Κύριε Πρίμπε. Είστε ο πρώτος που πρέπει να αποχωρήσει από την αίθουσα, επομένως μπορείτε να ξεκινήσετε εσείς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω ακόμη 42 λεπτά μέχρι την αναχώρηση του τρένου Έχω λίγο χρόνο. Όπως είπα, με πολύ μεγάλη προσοχή και εις βάθος εξετάζουμε την υλοποίηση της εκθέσεως και στη δεύτερη αναθεώρηση. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια, γιατί μας βοηθούν πολύ. Δεν συνηθίζουμε να είμαστε ε, καλοί και στοργικοί προς τους Αμερικανούς κοιτάμε πολύ μεγάλη προσοχή και από την πρώτη αναθεώρηση πρέπει να υπενθυμίσω ότι οι παρατηρήσεις σας είχαν βοηθήσει στον να εξασφαλιστούν βελτιώσεις και επίσης στη διαδικασία ελέγχου νομίζω ότι και αυτή συνέβαλε. Πρέπει να πω το άρθρο 4 όπως έχει συνταχθεί, όπως προέκυψε μετά τις πραγματεύσεις, έχει ως το δυνατόν πιο στενό πεδίο εφαρμογής. Φυσικά αυτό πάντοτε οδηγεί σε συγκρούσεις και συζητήσεις με τους Αμερικανούς και προσπαθούμε να τους πείσουμε να έρθουν πιο κοντά στις δικές μας θέσεις από το παρελθόν. Πάντως, ο μηχανισμός ελέγχου λειτουργεί και θα εξακολουθήσει να λειτουργεί. Ευχαριστώ την κυρία Σίπλ για τα συγχαρητήρια σε ένα βαθμό. Βεβαίως ακούσαμε τις προτάσεις σας, εισακούσαμε τις προτάσεις σας, αλλά πρέπει και εσείς να αντιληφθείτε ότι δεν έχουμε αρκετό προσωπικό λόγο και των περικοπών. Είναι πολύ δύσκολο για μας, είναι τεράστια επένδυση του να αποστείλουμε ακόμη έναν ε, υπάλληλο στη Washington. Τα καταφέραμε πάντως. Και χρειάστηκε και πολλή προσπάθεια για να πείσουμε τους Αμερικανούς να το δεχθούν, γιατί δεν είχαν τέτοια διάθεση. Δεν συνηθίζω να δίνω υποσχέσεις όταν δεν είμαι σίγουρος ε, για την έκβασή τους. Θα επανέλθουμε πάντως. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε η ίδια υποσχεθεί σύστημα οικονομικού εντοπισμού τρομοκρατών. Θα το κοιτάξουμε πάντως αυτό που είπατε. Θα σας ενημερώσουμε και πάλι το φθινόπωρο για την εξέλιξη στη μελέτη της υπόθεσης. Κυρία Κρούς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας και για τα σχόλιά σας. Αυτός ο δεύτερος έλεγχος ε, αφορούσε τη συμφωνία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τη στιγμή που η συμφωνία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε με βάση τις δικές μας αρμοδιότητες τήρησης του δικαίου το, το σημείο 2 του άρθρου 4 προβλέπει κάποιους όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις για το πώς θα πρέπει τα δεδομένα να μεταβάζονται προς οι ΗΠΑ. Και η κοινή εποπτική αρχή της Europol ε, έλεγξε την εφαρμογή αυτού του σημείου σε σχέση με το ρόλο που έχει η Europol ως προς το σημείο αυτό. Σε ό,τι αφορά το εδάφιο Α, το, το εδάφιο 2 του άρθρου 4, που λέει ότι το αίτημα των ΗΠΑ θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια όσο πιο σαφώς γίνεται τα δεδομένα που πρέπει να μεταβιβάζονται. Θα πρέπει να τεκμηριώνει σαφώς, προστίθεται το σαφώς. Θα πρέπει να τεκμηριώνει σαφώς το αίτημα σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα των στοιχείων. Επίσης, το αίτημα αυτό θα πρέπει να διατυπώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζει τον αριθμό των μεταβιβάσιμων στοιχείων. Και έτσι εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συμφωνία και θα πρέπει η κοινή Αποπτική αρχή να εξακριβώνει την ε, ε, εφαρμογή αυτού του άρθρου. Και εμείς στην έκθεση λέμε ότι η τεκμηρίωση εξακολουθεί να είναι αόριστη και όχι σαφής. Το ε, πεδίο εφαρμογή των ετοιμάτων εξακολουθεί να είναι αόριστο και γενικό και καλύπτουν ολόκληρο το χρόνο. Βέβαια, το είδος των πληροφοριών μειώθηκε που σημαίνει ότι όντως διαβιβάζονται λιγότερες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά έχουμε πληροφορίες που είναι ασαφείς, σχετικά αόριστες, δεν αφορούν συγκεκριμένα αιτήματα και δεν έχουμε στοιχεία για όλες τις κατηγορίες των ετοιμάτων, οπότε θεωρούμε ότι δεν έχουμε ε, μεταβίβαση του ελάχιστου αριθμού στοιχείων όπως απαιτείται από τη συμφωνία, αλλά περισσότερων στοιχείων. Γι' αυτό και εκφράσαμε ανησυχίε στην έκθεση. Πάντως συνεχίζουμε τις ε, εργασίες με την Europol και είχαμε πολύ αποτελεσματική και επικοδομητική συνεργασία. Προσπαθούμε να δούμε τι προσπάθειες απαιτούνται, τι νέα βήματα θα πρέπει να γίνουν ώστε να μπορέσει η Europol να εφαρμόσει αποτελεσματικά αυτό που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιλαμβάνεται στο εδάφιο 2 του άρθρου 4 της Συμφωνίας. Ευχαριστώ κύριε Ράιτ, ήρθε η σειρά σας. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αποτελεί απόδειξη των διαφορετικών ερμηνεών που δίνονται στις διαφορετικές τοποθετήσεις η συζήτηση που έλαβε χώρα. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 4. Άκουσα εκατό διαφορετικές εκδοχές του πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται το άρθρο 4. Ουσιαστικά η ε, Europol είναι αυτή η οποία έχει την άχαρη, το άχαρο καθήκον ε, να αποφασίζει τελικά αφού ακούσει όλες τις απόψεις και ε, θέσεις να εφαρμόζει το άρθρο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν, μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνάψει την συμφωνία αυτή και εμείς έχουμε αναλάβει την εφαρμογή της. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή, αλλά εν τέλει πρέπει να βρούμε και τον τρόπο υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των διασφαλιστικών δικλείδων. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε και πιστεύω ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά. Και από τα workshops που είχαμε με τις ΗΠΑ ε, και την GSP, και όλα τα μέλη είχαν την ευκαιρία να συστήσουν λεπτομέρως ε, στην πράξη, στην πραγματικότητα τι σημαίνει η προστασία και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και κάθε συγκεκριμένος πρακτικός τρόπος, ρεαλιστικός τρόπος βελτίωσης ε, της συμφωνίας ε, έχει εξεταστεί, τον έχουμε ε, συζητήσει και τον έχουμε εφαρμόσει. Περισσότερο από αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Όσον αφορά την πρόσβαση στην απόρριτη έκθεση, έχει χαρακτηριστεί η έκθεση αυτή ως απόρριτη, κατά Αιτήματος των Πολιτειών. Σωστή πιστεύω είναι η ε, ταξινόμηση αυτή ως απορρίτου. Ό,τι και να πει η JSP. Και εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αμφισβητήσω αυτό το, αυτή την ταξινόμηση. Αυτό το λέω όχι για να προτείνω μια παρελκυστική λύση, ούτε για να αποφύγω να δώσω απαντήσεις, απλώς γιατί θεωρώ ότι είναι το πιο σωστό να είναι ε, απόρριτα στοιχεία τα οποία εάν αποκαλυφθούν μπορεί να βλάψουν κάποιες επιχειρήσεις. Όταν έρθει η ώρα θα ενημερωθείτε. Thank you, ενδιαφέρον να ακούσουμε μια πιο λεπτομερή απάντηση του κυρίου Wainwright στις ερωτήσεις που τέθηκαν, ιδιαίτερα στην παράγραφο ε, στην οποία αναφέρθηκα, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα αυτά και ότι η συμφωνία αυτή σε αυτή την περίπτωση δεν έχει καμία αξία. Αυτό είναι περίεργο συμπέρασμα. Εγώ δεν θέλω να μας πείτε το τι έχει γίνει για να βελτιωθεί η εφαρμογή της συμφωνίας. Θα ήθελα τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Αυτά τα συμπεράσματα λοιπόν είναι ιδιαιτέρως ε, ανησυχητικά. Έχουμε ξεφύγει χρονικά. Περιμένουμε το επόμενο να συζητήσουμε, αλλά ένα λεπτό παρακαλώ για να δώσετε μια απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα που τέθηκε. Υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί περιορισμοί στον εντοπισμό και τη μετάδοση των πληροφοριών και δεδομένων. Κάποια ας πούμε δεδομένα δεν μεταδίδονται. Δεν παρακολουθούμε φυσικά όλες τις συναλλαγές στον κόσμο. Ένας πολύ μικρός ποσοστό, κάτω του 20% των οικονομικών συναλλαγών συμπεριλαμβάνονται και καλύπτονται από τη συμφωνία αυτή. Υπάρχουν λοιπόν περιορισμοί στην εντολή την σχετική με τον έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών. Καλώς σας ευχαριστώ. Ήταν μια πραγματική ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους όσους πήραν μέρος στη συζήτηση. Ευχαριστούμε εδώ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο κ. Σίφερ ήταν εδώ εκτός από τον κ. Πρίμπε. Κύριε Κρούς, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, κύριε Wainwright. Καλή επιτυχία. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Κάτι το οποίο δεν είναι άσχετο, είναι το 19. Η καζόμενη μεταφορά φυλακισμένων από πλευρά τη CIA. Η συγγήτρια είναι η κυρία Φλότρο.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 Calling for your attention and moving. We are here to consider the amendments of the draft. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες της ε, πρότασης την οποία συνέταξε η συνάδελφος κυρία Φλότρα. Detention and illegal detention of prisoners in European... Η καζόμενη μεταφορά φυλακισμένων από πλευρά της CIA. Η πρώτη σύνταξη της έκθεσης, εξέταση μάλλον της έκθεσης έγινε στην Λίμπε μετά στην ΑΦΕΤ, σύμφωνα με το άρθρο 50, η ψηφοφορία, η ψηφοφορία στη ΛΥΜΠΕ θα γίνει στην συνεδρίασή μας της 9ης και 10ης Ιουλίου. Στην ΑΦΕΤ η ψηφοφορία θα γίνει 15 Ιουλίου και όχι 25 Ιουνίου όπως είχαν στην αρχή προγραμματίσει. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Ελέν Φλότ πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τις τροπολογίες. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στην αντιπροσωπεία η οποία πήγε στο Βίλνιους της Λιθουανίας από τις 25 μέχρι τις 27 Απριλίου. Είχα την τιμή να καθοδηγήσω αυτήν την αντιπροσωπεία στην οποία συμμετείχε η κυρία Στίφλερ, η κυρία Φαγιόν, η κυρία Φλότρα, η κυρία Λάτφορντ και η κυρία Γκόμες. Λόγω απρόβλεπτων υποχρεώσεων η αντιπροσωπεία αυτή στη Λιθουανία αναγκάστηκα να φύγω εγώ στις 27 του μηνός και μετά η συγγήτρια κυρία Φλότρ ήταν υπεύθυνη για την αποστολή. Στόχος ήταν να κατανοήσουμε καλύτερα στη Λιθουανία τις δυσκολίες αυτή της συγκεκριμένης αποστολής η οποία ήθελε να προκαλέσει συζήτηση στα νέα στοιχεία για τα μυστικά προγράμματα κράτησης στην Λιθουανία και για τους μηχανισμούς διασφάλισης αποζημίωσης για τα θύματα, τα εμπόδια που συναντώνται και η βοήθεια την οποία μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγαμε επίσης και στη μυστική περιοχή, απόρριτη περιοχή του Ανταβίλιαε. Οργανώθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής εισαγγελίας με εκπροσώπους του Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το Προεδρείο της χώρας, με τους Υπουργούς Πολιτικής Αεροπορίας, Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας, Εξωτερικών Υποθέσεων τον Πρόεδρο του Βουλής και τον κύριο Αγκριμάτας Κλιούγκας, ο οποίος ήταν Γενικός Εισαγγελέας μέχρι το 2010 και ήταν υπεύθυνο για την υποδοχή της αντιπροσωπείας. Εμείς εκτιμήσαμε δεόντως την ετοιμότητα των λιθουανικών αρχών να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Αναγνωρίσαμε τις προσπάθειες έτσι ώστε να χυθεί φως σε αυτό το πρόγραμμα μεταφοράς κρατουμένων της CIA. Κάναμε συνεντεύξεις σε επίπεδο κοινοβουλευτικό και δικαστικό και να υπογραμμίσω και τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε ο πρόεδρος της Λιθουανίας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς ζητήσαμε όμως περιτέρω, περαιτέρω εξηγήσει σχετικά με τον περιορισμένο εύρος και το κλείσιμο της εισαγγελική έρευνας. Υποτίθεται μας είπε ο βοηθός εισαγγελέα ότι κανένας δεν κρατήθηκε εκεί και ο ρόλος ε, της αρχής του ε, κρατικού μυστικού, αν θέλετε, απορρίτου, είναι κάτι το οποίο αφορά και τα επίπεδα ελέγχου των μη εμπορικών πτήσεων, αφορά την αδυναμία των θυμάτων να προσφύγουν σε δικαστικές διαδικασίες όσο έχει κλείσει η έρευνα. Εκτιμήσαμε πάντως και την διαθεσιμότητα της εισαγγελίας και της λιθουανικής πολιτικής αεροπορίας να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Μια επιστολή που ζητά περαιτέρω πληροφορίες ε, υπεγράφει από εμένα τον ίδιο και την εισηγήτρια απεστάλλει στο γραφείο το Ισαγγελέα τον Ιούνιο του 12 και η απάντηση θα μεταφερθεί στους συντονιστές της Επιτροπής μας. Δίνω το λόγο λοιπόν τώρα πλέον στην κυρία Φλότρα. Θα ήθελα να εκφράσω και την εκτίμησή μου για την υποδοχή μας από πλευρά των λιθουανικών αρχών που θέλησαν να συνεργαστούν μαζί μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Προσπάθησα να ενσωματώσω τις βασικές πλευρές της επίσκεψής μας, τις νέες τροπολογίες και προσπάθησα να μεταφέρω στους συναδέλφους ότι έχουμε ακριβώς τη διάθεσή τους στην επιστολή που αποστήλαμε από κοινού με τον πρόεδρο στον Γενικό Εισαγγελέα. Μας είχε ζητήσει επίσημα επιτόπου για να μας δώσει πιο συγκεκριμένα έγγραφα και πιο απόρριτα μόνο εφόσον το ζητούσαμε γραπτά. Το κάναμε αυτό, δεν πήραμε ακόμα απάντηση Δεν αποκλείουμε να έλθουν ξεκάθαρες απαντήσεις σε ορισμένα θέματα, κάτι το οποίο θα μπορούσε σε συμφωνία με τους ε, σκιώδεις εισηγητές να οδηγήσει στην προσθήκη κάποιων παραγράφων στην έκθεσή μας. Αναφερθήκατε λοιπόν στο βασικό θέμα το οποίο είχαμε να αντιμετωπίσουμε ότι παρά τις δύο έρευνες στην Λιθουανία όλες οι ερωτήσεις δεν έτυχαν απάντησης από τότε και με το Eurocontrol και με την ανάλυση των πτήσεων έχουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες οι οποίες είναι ουσιαστικά κίνητρα για τον εισαγγελέα να ανοίξει εκ νέου μία προκαταρκτική έρευνα. Πόσο μάλλον που εξέφρασε και την επιθυμία του να παραμείνει δεκτικός στην δυνατότητα μιας νέας έρευνας. Εκεί βρισκόμαστε τώρα με τη Λιθουανία. Η αντιπροσωπεία αυτή ήταν χρήσιμη θα έλεγα. Ε, με την εμπειρία που πήραμε θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε το κείμενο με τις τροπολογίες. Τώρα να έλθω στις υπόλοιπες τροπολογίες είναι 143. Ομολογώ ότι 22 από αυτές προέρχονται από εμένα. Και αυτές οι 22 ακριβώς κάνουν αυτό το οποίο είπα. Καλύπτουν δηλαδή τις πρόσφατες αναλύσεις, τις πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις τις οποίες μας έδωσαν οι υπηρεσίες του Eurocontrol και που περιλαμβάνουν σημαντικά στοιχεία για τη Ρουμανία και τη Λιθουανία. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες σε σχέση με την επίσκεψη που έκανα στις 16 Μαΐου στην Πολωνία, όπου συναντήθηκα με τη Γενική Εισαγγελία και κάποιες άλλες συζητήσεις και πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση στη Ρουμανία. Αυτά για τις 22 δικές μου τροπολογίες, μπορώ να επανέλθω. Πολλοί συνάδελφοι κατέθεσαν τροπολογίες οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές μπορώ να αναφερθώ στα θέματα πάνω στα οποία θα μπορέσουμε να κάνουμε συμβιβαστικές συζητήσεις, προτάσεις, συγγνώμη. Είναι τροπολογίες οι οποίες εγγράφονται, θα έλεγα, στην προβληματική της καταπολέμησης της τρομοκρατίας σε σύνδεση με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει το θέμα του ελέγχου των δραστηριοτήτων των μυστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως κοινοβουλευτικός έλεγχος. Πολλές τροπολογίες ε, ε, κατέθεσαν, κατετέθησαν και θα οδηγήσουν σε μια συμβιβαστική τροπολογία. Πολλοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνεται καταχρηστική χρήση του κρατικού απορρίτου και δεν θα πρέπει να είναι ένα άλοθη για την ε, πιθανή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ορισμένε τροπολογίες σε κάποια προληπτικά μέτρα για το μέλλον, την αξιολόγηση των πρακτικών κτλ. Είναι κάποιες πιο γενικές τροπολογίες στα πλαίσια της πολιτικής καταπολέμησης της τρομοκρατίας και κάποιες από τις τροπολογίες αυτές μπορούν κάλλιστα νομίζω να γίνουν δεκτές γιατί θα πυκνώσουν και θα πλουτίσουν το κείμενο. Θα ήθελα να σας προτείνω επίσης να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε κάποια συγκεκριμένα θέματα για να μπορέσουμε να κάνουμε και συγκεκριμένες ε, επιλογές. Ότι αναφέρεται στο παρελθόν να συμπεριληφθεί στις αιτιολογικές εκθέσεις, την αιτιολογική μάλλον έκθεση, και να προσπαθήσουμε να, να περιοριστούμε στις συστάσεις σε ό,τι σε επίπεδο επικαιρότητα θα έλεγα εξηγεί τις πολιτικές κινήσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν και τις οποίες μπορούμε να συμπεριλάβουμε στην έκθεση για το παρόν και το μέλλον. θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το τι ε, πράγματι είναι ουσιαστικό στην έκθεση αυτή ε, το περιεχόμενο δηλαδή των ερευνών, των ανακρίσεων που έχουν γίνει σχετικά με τις δράσεις των κρατών μελών σε σχέση με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Βέβαια δεν υπάρχει ισότητα, δεν υπάρχει μία παράγραφος για κάθε μία από 27 χώρες, τότε θα μιλούσαμε για ισότητα αλλά θα πρέπει να συνεννοηθούμε εδώ. Έχουμε να κάνουμε ότι αυτό που έχει σημασία είναι η ε, τόπη κράτησης και οι μετακινήσεις των κρατουμένων. Γιατί αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Οι πτήσεις στις οποίες μπορούμε να αναφερθούμε είναι ενδιαφέρουσες παρά μόνο μέσα σε αυτή την προοπτική. Στον βαθμό που συνδέονται δηλαδή με τη μεταφορά κρατουμένων σε μυστικούς τόπους κράτησης. Ταυτόχρονα και σε σχέση με τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είτε δικαστικές είτε κοινοβουλευτικές, όχι μόνο να τις αναφέρουμε, αλλά να αναφερθούμε συγκεκριμένα στα συμπεράσματά τους. Πολλές τροπολογίες, σαν παράδειγμα, προτείνουν πάνω στην ε, συγκεκριμένη έκθεση. Εν πάση τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έκθεσης ε, λέγεται ότι δεν έχει αποδειχθεί κάτι, οπότε δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι κάτι συνέβη. Αυτή είναι η θέση η οποία είναι περίπου η επίσημη θέση των Ρωμανικών αρχών και η οποία θα έλεγα προσπαθεί να επανέλθει στην έκθεσή μας με 60 τροπολογίες αυτό εξηγείται από την κατάσταση στη Ρουμανία, πρέπει να πούμε το τι συνέβη. Δεν θα πρέπει όμως εμείς να μην ονοματίσουμε αν θέλετε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες, καταστάσεις και έρευνες οι οποίες είναι τέτοιας φύσεως που θα δικαιολογούσαν την νέα έρευνα, μια πιθανή νέα έρευνα η έκθεση καλό θα είναι να το πει αυτό. Εάν δεν το κάνει φοβάμαι ότι δεν θα παρουσιάζει περιεχόμενο, αξιοπιστία και ενδιαφέρον. Έρχομαι τώρα στις συμβιβαστικές προτάσεις, οι οποίες θα είναι στη διάθεσή σας την επόμενη εβδομάδα. Είναι σαφές ότι επί της παραγράφου 1 χωρίς πολλές δυσκολίες και όπως είπα προς την κυρία Στρίφλερ και την κυρία Σταντζόν μπορούμε να πούμε ότι τα κράτη δεν θέλουν συστηματικά να μη σέβονται νόμο, αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν φέρει εις πέρας πάντα τις ε, αποστολές τους αυτές σωστά. Νομίζω ότι μέσω αντικατάστασης μια τροπολογίας από κάποια άλλη μπορούμε να καταλήξουμε σε διατυπώσεις που θα ικανοποιήσουν τους συναδέλφους διευκρινίζοντας την παράγραφο 1. Για την παράγραφο 2 Δεν υπάρχουν πολλές τροπολογίες στην παράγραφο 2. Προτείνω προς την κυρία Στρίφλερ να θεωρήσει την 66, τροπολογία της 66 σαν προσθήκη. Να πούμε ότι κάποιες χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη διεξαγωγή των ερευνών <clears throat> και παράλληλα με τις δυσκολίες αυτές έχουμε πλέον ελλείψεις στην πληροφόρησή μας κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο την αμοιβαία αξιοπιστία μας. Επί της παραγράφου 3... Ε, δεν έχω τίποτα ούτε για την παράγραφο 4. Τώρα για την παράγραφο 5. Oui, qui concerne donc... Euh, η παράγραφος αυτή λέει ότι οι έρευνες θα πρέπει να στραφούν γύρω από τις μυστικές φυλακές και τους ε, πιθανούς ε, κυκρατουμένους. Νομίζω ότι έχουμε εμπνευστεί από τις ε, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξού και οι, οι τροπολογίες 82, 83, 84, Βερζιά και Κουέλιο που θα μπορούσαν κάλλιστα να συνδυαστούν σε μια συμβαστική λύση. Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 6, ε, ερχόμαστε εδώ στο θέμα της Ρουμανίας. Μιλήσαμε για το θέμα της Ρουμανίας. Ε, κυρία Σλίφερ κατέθεσε τροπολογία. Θα ήθελα η μνήμα της σχετικής έρευνας να γίνει στην αιτιολογική έκθεση. Και εδώ να απευθύνουμε έκκληση στις δικαστικές αρχές να ξεκινήσουν ανεξάρτητη έρευνα με βάση νέα στοιχεία για τις πτήσεις μεταξύ Λιθουανίας και Ρουμανίας. Μάλιστα, έχουμε από την τελευταία ανάλυση των στοιχείων της Eurocontrol νέα στοιχεία που τα παρουσίασε και στη συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών. Σε ό,τι αφορά τη Λιθουανία τώρα, νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε με τις κυρίες Βερζιά και Σίφλερ που κατέθεσαν τροπολογίες. Μάλιστα η κυρία Σίφλερ κατέθεσε τις τροπολογίες 99, ε, 100 και 101. Στην 101 ε, επαναλαμβάνεται αυτό που είπαν ε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν ε, παραβιάστηκε η κυριαρχία, η εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Το είπαν και για τη Λιθουανία και γενικώ. Πιστεύω ότι στην τροπολογία αυτή για τη Λιθουανία και ε, τις δηλώσεις των ε, Αμερικανικών αρχών να τις αναφέρουμε στις ε, αιτιολογικές σκέψεις. Εκεί που μιλάμε για τις δηλώσεις της κυρίας Κοντολίτσα Ράης και εκεί που μιλάμε γενικά για τις δηλώσεις που έγιναν όχι μόνο για τη Λιθουανία. Θα προτείνω συμβεστική τροπολογία για την παράγραφο 10 που μιλά για τα δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες. Μερικές χώρες δεν έχουν δώσει ακριβείς πληροφορίες. Ούτε δημοσίευσαν ε, τις ε, πληροφορίες για τις πτήσεις που ενδεχομένω γίνονταν με συμμετοχή της CIA. Αναφέρονται πολλές χώρες. Θα έλεγα να πάρουμε τον πιο περιεκτικό κατάλογο των χωρών, του κυρίου Κοέλιο δηλαδή, και να δούμε πώς θα συμπεριλάβουμε και το δικαίωμα πρόσβασης και το θέμα των απαντήσεων που δεν δόθηκαν. Αυτά θα τα αναφέρω στη συμβιβαστική τροπολογία. Στη συνέχεια, περνάμε στην παράγραφο με τις πολιτικές πρωτοβουλίες που θα θέλαμε να ληφθούν από το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο στις τακτικές συνεδριάσεις που γίνονται ε, με τα Εθνικά Κοινοβούλια, ώστε να προχωρήσουμε και στις έρευνές μας αλλά και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς των δραστηριοτήτων των μυστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ασφάλειας. Ως προς το Συμβούλιο... Α, υπάρχει μια σειρά τροπολογιών όπου αναφέρεται το θέμα τι θα ζητήσουμε από το Συμβούλιο. Θα ζητήσουμε να αναγνωριστεί η ανάμειξη του, να ζητήσει δημοσίου συγγνώμη, να αναγνωρίσει τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Ας αφήσουμε τις ε, συγγνώμες και τις δικαιολογίες, γιατί ίσως είναι περίπλοκο αυτό το θέμα και ποιος θα κάνει τη σχετική δήλωση. Πάντως, να αναγνωριστεί ε, με κάποιο τρόπο η ανάμειξη του Συμβουλίου και των κρατών μελών στην υπόθεση αυτή και να αναφερθούν οι δυσκολίες για την ενημέρωση του συστήματος και της ε, ε, ανάμειξη και το θέμα της διαλέγκας από τη δικαιοσύνη. Θα μπορούσα λοιπόν να σας υποβάλω εδώ μια συμβαστική τροπολογία. Δεν ξέρω ποιος είχε καταθέσει αρχικά τροπολογίες. Α, οι κύριες Σίφλερ και Βερζιά για την παράγραφο 11 ως προς τη συμμετοχή του Συμβουλίου. Δεν θα αναφερθώ λεπτομεριακά στις 143 τροπολογίες, γιατί πολλές από αυτές αναφέρονται σε ένα θέμα που εγώ είχα παραλείψει, αλλά τελικά θα το προσθέσω και θα το συνδυάσω με κάτι άλλο, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των πτήσεων και τον έλεγχο των αεροσκαφών. Το θέμα της αναθεώρησης της ε, σύμβασης ε, του Σικάγου, για παράδειγμα, ε, είναι θέμα που υπέβαλα στις τροπολογίες τους η κυρία Γκόμες και ο κύριος Κοέλιο. Νομίζω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τις δύο τροπολογίες και να προσθέσουμε μία αναφορά και στο σημείο αυτό. Δεν, ξέρω, δεν ξέρω αν πρέπει να το συνδέσουμε με το θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Θα δω τι τελική μορφή θα έχει έκθεση. Πάντως, ήδη αρχίζει να προδιαγράφονται οι, οι βασικές ε, γραμμές της οριστικής πια μορφή της έκθεσης μετά από τις τροπολογίες που υποβάλλατε και τις συμβαστικές τροπολογίες που θα σας υποβάλλω την επόμενη εβδομάδα. Ήδη έχουμε προγραμματίσει συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών στο Στρασβούργο για την 5η Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το επιβεβαιώνει η γραμματεία. 5 Ιουλίου συνεδρίαση με τους σκιώδες εισηγητές. Και αυτά ήταν τα πιο βασικά στοιχεία της έκθεσης. Αν κάτι παρέλειψα θα μου το επισημάνετε φαντάζομαι και περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Φλότρ για την παρουσίαση των εκθέσεων για την επίσκεψη της αντιπροσωπής στη Λιθουανία. Και τώρα, ώρα για συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένο και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φλότρο για την θέση της εδώ. Ελπίζω να κάνει δεκτές τις τροπολογίες που καταθέσαμε. Ίσως ε, να προτείνει και συμβαστικές τροπολογίες. ήθελα να τοποθετηθώ προς τις ε, τροπολογίες και να εξηγήσω γιατί τις κατέθεσα. Καταρχάς, στόχος των ε, τροπολογιών. Για μένα τουλάχιστον ήταν να προσεγγίσουμε το πεδίο της πραγματικότητας περισσότερο και να αποφύγουμε τις ε, μη εμπεριστατωμένες δηλώσεις. Η προστασία των δικαιωμάτων είναι ένα τόσο σημαντικό θέμα που δεν πρέπει να ε, βάλουμε κατά άλλων χωρίς να, έχουμε, να μπορούμε να στηριζόμαστε σε στοιχεία. Η πενιγμή λοιπόν για παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων στηριζόμενη μόνο στα δημοσιεύματα του τύπου είναι μάλλον επικίνδυνη. Με τις τροπολογίες μου λοιπόν επιδιώκω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι οι μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιήσει τα κράτη-μέλη για να διαφωτίσουν αυτές τις ε, μεταφορές κρατουμένων ε, σε μυστικές ε, ε, φυλακές ήταν διαφορετικές. Άλλα κράτη θέσπισαν ε, εξεταστικές επιτροπές, άλλα λιγότερο ε, εμφανείς διαδικασίες κτλ. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Ρουμανία έγινε έρευνα από το Κοινοβούλιο το 2008. Στην, στο σχέδιο εκθέσεων όμως δυστυχώ δεν αναφέρεται καθόλου αυτό το γεγονός. Εγώ προσωπικώς πιστεύω ότι ένα Εθνικό Κοινοβούλιο, όπως βέβαια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, αξίζει του σεβασμού μας και της προσεκτικής εξέτασης της δράσεώς του πλευράς μας. Εάν βεβαίως υπάρχουν ε, αποδεικτικά στοιχεία για την ε, παραβίαση των προδικαιωμάτων θα πρέπει να εξεταστούν όπως ορίζουν οι εθνικοί και οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Πάνω απ' όλα όμω, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όσο και είναι ρόλο μα να προστατεύουμε το ευρωπαϊκό συμφέρον δεν μπορούμε να υποκαθιστούμε τι κριτικές αρχέ ούτε να ανατρέπουμε τη σχέση ε, με τον νόμο του, την υποχρέωση σεβασμού στον νόμο δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Νσιού. Κυρία Ινφέλτ έχει το λόγο. Πρόεδρε ευχαριστώ. Φαίνεται ότι η φωνή μου δεν έχει βελτιωθεί παραμένω βραχνή. Θα ήθελα πολύ στο να απαντήσω στον ε, συνάδελφο κύριο Ενσού, λέγοντα ότι πολλέ είναι τροπολογίε που υπηρετήσαν, αλλά θα προτείνω να μην υποστηρίξουμε καμία ρουμανική τροπολογία. Νομίζω ότι είναι κάπω δύσκολη θέση μα όταν συζητούμε για τόσο σημαντικού ε, και σοβαρού υπενιγμού που έχουν μεταφέρει όχι μόνο τα μέσα μαζική ενημέρωση, γιατί εμεί το θέμα αυτό το παρακολουθούμε τόσα χρόνια. Και βεβαίω έχετε κάθε δικαίωμα. Είναι πολιτική η έρευνα και όχι ε, δικαστική. Δεν είμαστε δικαστήριο, δεν πρέπει να αποδείξουμε κάθε μεμονωμένο περιστατικό. Αλλά δεν μπορείτε να αρνηθείτε την ύπαρξη όλων αυτών των στοιχείων, ως βουνού αποδεικτικών στοιχείων για όλα αυτά τα περιστατικά που έλαβαν χώρα σε σχέση με μία χώρα. Δεν μπορείτε να μας ότι δεν έχουν καμία ε, σχέση. Σημασία έχει, και σε αυτό πρέπει να καλέσουμε σε λογοδοσία τους υπέτειους, η ευρωπαϊκή, το ότι η ευρωπαϊκή οικογένεια, τα ευρωπαϊκά κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέπραξε είναι συνένοχος σε παραβίαση των Το να οφείλεται αυτό στην επιλογή της κυβέρνησης της χώρας που εκπροσωπείτε εσείς ή εγώ δεν έχει σημασία και χωρίς να είναι η δική μου χώρα τόσο πολύ στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ε, είμαι, θεωρώ προτιμότερο, εάν υπάρχουν κάποιοι πενιογμοί, έστω και λίγοι και ισχνοί, να διερευνηθούν διεξοδικά και θα αισθάνομαι καλύτερα για την πατρίδα μου, εάν ξέρω ότι έχουν εξεταστεί όλα και δεν πρόκειται να επαναληφθεί τίποτα τέτοιο. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με την ε, ηθική ακερότητα της Ευρώπης στο σύνολό της όχι μόνο για τη Ρουμανία, όχι μόνο για, τη ε, για την Ολλανδία, αλλά για τις κατοχώρες, αλλά για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία και όλα τα κράτη. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί θα πρέπει να επιδιώκουμε την απαλήψη μιας αναφοράς σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, γιατί το θέμα δεν αφορά κράτη-μέλη, αλλά τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα. Και κάτι άλλο το οποίο είχα επισημάνει και στη συζήτησή μας στο Στρασβούργο τελευταία φορά στρατηγική σημασία ε, παρατήρηση, στρατηγική φύσεω. Μιλούμε για γεγονότα, για υπενιγμού, ε, για ισχυρισμού, χωρί όμω να έχουμε συγκεκριμένη εικόνα για το τι συνέβη. Τι θα γίνει λοιπόν αυτή την έκθεση. Τα κράτη-μέλη έχουν ε, αγνοήσει την προηγούμενη έκθεση, ούτε καν τα ενδιαφέρει αυτή η έκθεση. Και από εδώ που κάθομαι, αγαπητοί φίλοι, βλέπω ότι στα δεξιά τη αίθουσα δεν κάθεται κανένα. Πού είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Α, μάλιστα, είναι εκπρόσωπο, μάλιστα από το γραφείο του ΕΛΚ, από το προσωπικό δηλαδή. Γεια σου Μάικλ. Αλλά πού είναι οι βουλευτέ, Μιλούμε για Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα, παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων, παραβίαση του διεθνού δικαίου πάνω σε ευρωπαϊκό έδαφο Και γιατί αυτό θεωρείται ω ίσονο σημασία σύντομα που θα πρέπει να συζητήσει μόνο η συγγήτρια ε, και μια χούφτα σκιώδης συγγητές, στους οποίους δεν συγκαταλέγεται καν ο σκιώδης του ΕΛΚ. Το θέμα βέβαια συζητούμε το τι μπορεί να συνέβη, τι μπορεί να μην έχει συμβεί, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι κάποιοι Ευρωπαίοι αρνούνται τα γεγονότα, αρνούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Και αυτό το αποδεικνύουμε την αποσία του ορισμένη. Εμεί οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή κοινωνία αρνούμεθα να έρθουμε αντιμέτωποι με τα εγκλήματα που στο όνομά μα έχουν διαπραχθεί. Ναι, κυρία Λάτφορτ, και εσεί, κύριε Ένσιου, θα σα δώσω το λόγο, αλλά α ακούσω πρώτα τι έχει να πει η κυρία Λάτφορτ και μετά θα γυρίσουμε σε εσά. Η κυρία Λάτφορτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ως σκιώδη συγκήτρια το... της ομάδας μου, αλλά και ως ε, συντάξει γνωμοδότηση εκ μέρου τη ΑΦΕΤ, λαμβάνω τον λόγο. Δεν θέλω να πω ότι ναι, παρακολουθώ μεγάλη προσοχή το όσα είπε η κυρία Νετφέλντ. Πολλά έχουμε να πούμε. Η κυρία Φλότρη με βεβαία θέλει να έχει μια προσέγγιση προσεκτική και λογική. Επιδεικνύει ευαισθησία. Θα ήθελα ωστόσο να πω ότι από τα όσα μπορούμε να διαπιστώσουμε δεν αποδεικνύεται πουθενά ότι υπήρξε συστηματική παράδοση, κράτηση, παράνομη μεταφορά κρατουμένων δεν έχει ακόμη ε, διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κράτος μέλος το οποίο μέχρι τώρα να έχει δώσει επαρκείς εξηγήσει για, τις, ε, για τους ισχυρισμού, είτε πρόκειται για ΜΜΕ, είτε πρόκειται για μη κυβερνητικέ οργανώσεις, είτε πρόκειται για πρώην ε, πράκτορες της CIA δεν βλέπω να πληρούνται, να, ε, να αποδεικνύονται τα όσα έχουν ε, υποθεί. Επίσης θα ήθελα να πω ότι όταν ξεκίνησε η ιστορία με την παρακολούθηση των υποκλοπών τηλεφώνων στο Ηνωμένο Βασίλειο με την υπόθεση Λόρινσον, αυτή ξεκίνησε όχι γιατί η αστυνομία είχε διερευνήσει. Του αντίον μα, επειδή η αστυνομία δεν είχε παρκώ διερευνήσει τι τηλεφωνικέ υποκλοπέ και έτσι ξεκίνησε η εφημερίδα Guardian. Άρα έχουμε αυτό τον, ε, την δημοσιογραφία, τη λεγόμενη ερευνητική, η οποία πολλές φορές έχει ξεκινήσει τέτοια, τέτοια θέματα που οδηγούν τελικά σε απόδειξη εγκλημάτων, όπως είχαμε και στις ΗΠΑ με την Washington Post και τη Stuxnet και όλες τις ε, κυβερνοεπιθέσεις, που έχουν ε, σε ένα βαθμό αποδειχθεί. Περιμένουμε να δούμε αν πλήρως θα ε, ελεγχθούν όλα αυτά. Επομένως, πρέπει να έχουμε έναν ισορροπημένο, μια ισορροπημένη αντιμετώπιση, χωρίς να προσβάλλουμε καμία χώρα φυσικά και τις ευαισθησίες της, αλλά ζητώντας μια πλήρη δικαστική διερεύνηση Τη υπόθεση γιατί ε, οι βουλευτέ ε, τουλάχιστον στη δική μου την ένωμη τάξη, δεν θα μπορούσαν ε, να κάνουν μια πλήρη έρευνα μια υπόθεση. Μέχρι τώρα οι αντίστοιχε αρχέ στο αμένο Βασίλειο, παραδείγματι, λογοδοτούσαν μόνο στον Πρωθυπουργό. Οι αρμόδιε αρχέ, οι Υπηρεσία πληροφοριών δηλαδή. Και έτσι οι βουλευτέ δεν είχαν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Άρα, ναι, θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να μην ενοχλήσουμε, να μην ε, ε, δημιουργήσουμε, να μην ταράξουμε τα νερά ε, και να μην ενοχλήσουμε ευαισθησίε μεν, αλλά πάλι πρέπει να κοιτάξουμε τι έχει πραγματικά συμβεί. Και συμφωνώ με την Σοφή ότι μας αφορά όλους αυτή η υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σύνολο κάποια κράτη-μέλη επέτρεψαν ή όλα τα κράτη-μέλη επέτρεψαν να συμβούν όλα αυτά, έστω και αν δεν έλαβαν χώρα πάνω στο εδάφο του αυτέ οι συλλέψεις ή μεταφορέ, έκλεισαν τα μάτια και δεν έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει, το έχω σημειώσει και στην γνωμοδότησή μου, θέλουμε περισσότερη υποστήριξη από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Ελπίζω και το ΕΛΚ και του συντηρητικού μεταρρυθμιστέ του Ηνωμένου Βασιλείου και το είχαμε δει άλλωστε και στην προηγούμενη έκθεση με το Γκουαντάνομο που είχε πάνω από 500 ψήφου υποστήριξη στην Ολομέλεια, δηλαδή είχε από όλα τα κόμματα υποστήριξη και έφερε κάποια αποτελέσματα ουσιαστικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των συνθήκων κράτηση στον Κουαντάνομο. Άλλαξε η ζωή των ανθρώπων αυτών ουσιαστικά. Λοιπόν, ναι, βεβαίω μπορούμε να δείξουμε μια κάποια κατανόηση και ευαισθησία, αλλά μέχρι ενό βαθμού. Προκειμένου να μπορέσουμε να ε, εξασφαλίσουμε σύμπραξη όλων των πλευρών, ναι, θα δείξουμε ευαισθησία, όχι όμως αδυναμία. Και για τον κύριο Ενσιού. Μα λέτε ότι δεν έχουμε αποδείξει γιατί δεν, έχει, ε, δεν υπάρχουν αποδείξει και έτσι δεν χρειάζεται να ξεκινήσει δικαστική διαδικασία. Μα το αντίστροφο ισχύει. Μόνο με βάση αποδείξει, μπορεί να, μόνο αν υπάρχουν αποδείξει μπορεί να προκύψει ε, ετοιμιγορία, δηλαδή βάση αποδείξεων, συλλέγοντας αποδείξεις αποφασίζουμε αν μπορεί να γίνει δικαστική διαδικασία και όχι το άλλο στην τροφό. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της απογευματινής συνεδρίασης. Θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Έντσιου βέβαια. Δεν χρειάζεται τώρα να ξανανοίξουμε όλη τη συζήτηση. Αλλά επειδή έγιναν προσωπικά σχόλια για σας, έχετε το λόγο να δευτερολογήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως έγινε κάποια παρανόηση των παρατηρήσεών μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι δεν είμαι κατά της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, είτε είναι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι πολίτες οποιασδήποτε άλλης χώρας του κόσμου. Εγώ καθ' όλη τη σταδιοδρομία μου και την πολιτική τάχθηκα υπέρ της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η κυρία Ιντβελτ μίλησε για απτές αποδείξεις που στοιχειοθετούν ε, και τεκμηρώνουν τους χειρισμούς. Πού βρίσκονται αυτές οι απτές αποδείξεις. Αν κάποιος έχει τεκμήρια να μας τα παρουσιάσει. Να απευθυνθεί στις ρουμανικές αρχές ε, ή στο Κοινοβούλιο, να δημιουργηθεί μια νέα ερευνητική επιτροπή και αν όντω ε, διαλευκανθεί η περίπτωση, αν όντως επαληθευτούν αυτές οι αποδείξεις να αναλυφθούν μέτρα και δράσεις κατά της Ρουμανίας. Έχουμε στην αίσθηση ότι έχουμε ξεπεράσει το πολιτικό επίπεδο και εμπλεκόμαστε σε δικαστικά θέματα που σίγουρα ξεφεύγουν από τις δικές μας αρμοδιότητες. Δεν μπορούμε εμείς ε, να ε, καταλήγουμε σε αποφάσεις μόνο και μόνο επειδή ένας δημοσιογράφος ε, ε, ξέδωσε άρθρο σε μια εφημερίδα και μετά να διαρριγνύουμε τα ημάτια μας για την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, γιατί θεωρούμε ως απαράβατη αλήθεια αυτά που διαβάσαμε σε μια εφημερίδα. Θα ήθελα επίσης ε, από την έκθεση να διαγραφεί σαφή σημειά συγκεκριμένων κρατών μελών. Γιατί αν εγώ ε, λεκιάζω την γραβάτα μου και προσπαθώ να την καθαρίσω, τελικά ο Λεκές δεν φεύγει, θα πρέπει να την πετάξω. Αλλά μένει ο Λεκές, καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και αν κατονομαστούν συγκεκριμένε χώρες στην έκθεση αυτή, ακόμη και αν αθωωθούν εκ των υστέρων, θα παραμείνει αυτή η μνήα και η κυλίδωση της φήμης τους. Θα ήθελα, κύριε Λάτφορτ, να σας πω ότι συμφωνώ μαζί σας, αλλά να σας κάνω μια ερώτηση. Αν μετά από μια δικαστική έρευνα και μια ανάκριση που γίνεται από τις αρμόδιες αρχές για τέτοιου έρευνα. αν μετά το πέρας της έρευνας διαπιστωθεί ότι οι δηλώσεις στον τύπο και τα άρθρα ήταν αναδαφικά, τι θα γίνει. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος δημοσιογράφος ε, γράφει ένα άρθρο είναι και γεμάτο με ακριβείς πληροφορίες. Κάτι τέτοιο περίπου συμβαίνει και στο ρωμανικό τύπο. Τι θα γίνει όμως αν δεν επαληθευτούν αυτές οι πληροφορίες μετά από τη δικαστική έρευνα. Εγώ είμαι υπέρ της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί ότι είχαμε τέτοιες περιπτώσεις στην ΑΒ χώρα. Να πούμε γενικά ότι ότι θα πρέπει να γίνουν έρευνες και αν υπάρξουν, συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία μετά από τη διερεύνηση, να τιμωρηθούν οι πέτοι με βάση το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, αλλά να μην στιγματίζουμε χώρες. Καλώς, σαφές ε, το σχόλιο σας κύριε Εντσίου. Θα δώσω τώρα το λόγο πάλι στη συγκεκριά μας για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Κυρία Φλότρ, ευχαριστώ. Κατανοώ τη θέση του συναδέλφου. Όντως υπάρχει μια μνήμα της κοινοβουλευτικής έρευνας που ξεκίνησε στη Ρουμανία, αλλά δεν αναφέρθηκαν τα πορίσματα αυτής της έρευνας. Αναφέρουμε στην ιδεολογική σκέψη ποιο ήταν και το πόρισμα αυτής της κοινοβουλευτικής έρευνας στη Ρουμανία. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπο που διεξήχθη αυτή η κοινοβουλευτική έρευνα, το κατά πόσο δημοσιεύθηκαν τα απορίσματα, τα σχετικά έγγραφα, όλα αυτά τα θέματα προκάλεσαν κριτικές επικρίσεις όχι μόνο από δημοσιογράφους. Αν κάποιος ενδιαφέρθηκε για το τι συνέβη στη Ρουμανία, διαπίστωσε ότι υπήρξαν πολλές παραλήψεις εκ μέρους των αρμόδιων αρχών και αυτό το επισήμαναν δημοσιογράφοι, αλλά η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστήριων, έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, έκθεση του κ. Μάρτη δεν ήταν, ήταν πολύ σοβαροί άνθρωποι που ισχυρίστηκαν της ελλείψης αυτής της έρευνας. Η Ρουμανία λέει το θέμα θεωρείται λήξαν, αλλά δεν ισχύει αυτό γιατί καθημερινά έχουμε νέες στοιχεία και νέες πληροφορίες. Συνεχίζονται έρευνες, συνεχίζονται δικαστήρια, υπάρχει κρεμή και η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και μάλιστα έγιναν εκκλήσεις σε υψηλό επίπεδο και από τα Ηνωμένα Έθνη και από το Συμβούλιο της Ευρώπης και διαβήματα προς τη Ρουμανία γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία που ε, θεμελιώνουν την ε, ανάγκη για νέα έρευνα. Έχετε δίκιο. Δεν πρόκειται εμεί να εξαγάγουμε αυτή την έρευνα. Δεν είναι δική μα αρμοδιότητα. Ούτε εμεί συγκεντρώνουμε τα νέα στοιχεία. Απλώ διαπιστώνουμε ότι έμειναν αναπάντητα κάποια ερωτήματα. Διαπιστώνουμε ότι οι έρευνε δεν ήταν και τόσο αξιόπιστε, διαφανεί, ευρυθεί και αποτελεσματικέ. Επίση, μπορούμε να ενθαρρύνουμε, και αυτό το στόχο έχει έκθεση, να ενθαρρύνουμε τα κρατημέλια, όχι να τα στιγματίσουμε. Το λέμε συνεχώ στην έκθεση. Και το λένε και, το είπαν και οι προλαλήσαντες, ότι το θέμα είναι ευρωπαϊκό. Το διακύβευμα είναι ευρωπαϊκό και η Ρουμανία θα πρέπει να συμβάλλει στην ε, πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την ανέβρεση της δικαιοσύνης και της αλήθειας. Και η Ρουμανία και η Λιθουανία και η Πολωνία και άλλες χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία. Οπότε αυτή η αρχή της αλληλεγγύης και της συνεργασίας καθώς και της υποχρέωσης που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαλευκάνει την υπόθεση, Μα οδήγησαν στο να απευθύνουμε έκκληση προ τη Ρουμανία να αναλάβει το τμήμα τη δική της ευθύνη. Υπάρχουν πολλά στοιχεία για του μυστικού τόπου κράτηση. Δεν είναι μόνο ένα δημοσιογράφο που θέλει να τις πάσει στη Ρουμανία, που θέλει να ενοχλήσει τι Ρουμανικέ αρχέ. Είναι υπερβολικό. Έγινε διασταύρωση πολλών πληροφοριών που κατέθεσαν πολύ σοβαροί οργανισμοί όπως ο Οργανισμός για την πρόληψη των βασανιστήριων. Ας μην εξετάζουμε λοιπόν επί επιπόλαια αυτά τα πράγματα. Εμείς φυσικά δεν μπορούμε να πούμε τι εστί απόδειξη και τι όχι. Γι' αυτό ζητούμε να γίνει έρευνα, για να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχουν αποδείξεις. Ούτε εσείς ούτε εγώ, από όπου και αν καταγόμαστε, δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε κάτι τέτοιο. Η έρευνα θα δείξει αν υπάρχουν αποδείξεις. Γι' αυτό και ζητούμε τη διεξαγωγή έρευνας έχουν κατατεθεί περίπου 60 τροπολογίες με αυτό το περιεχόμενο πάνω κάτω. Δηλαδή προσπαθούν να αποδυναμώσουν, να μην αναγνωρίσουν, να παραλείψουν, να θεωρήσουν ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε και το θέμα έληξε. Όχι, αλλά αυτό είναι μια άρνηση της πραγματικότητας. Ε, εθελοτυφλία ε, απέναντι στην κατάσταση και άρνηση της ανάληψης ευθύνης. Είμαι πρόθυμη να συζητήσω με τους συντάκτες των τροπολογιών, αλλά όχι με τη βάση που προτείνετε εσείς. Γιατί νομίζω ότι έτσι δεν θα μας πάρουν στα σοβαρά. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάει για τέτοια θέματα θα πρέπει να είναι αξιόπιστο, αξιοσέβαστο και να υποβάλει συστάσεις που θα ε, δώσουν μια όθηση. Και για την περίπτωση της Ρουμανίας πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε μια όθηση. Και όσο πιο γρήγορα κινητοποιηθούν οι ρωμανικές αρχές, τόσο το καλύτερο γιατί αν η Λιθουανία ξανανοίξει, ξαναρχίσει η έρευνα, είχαμε τα τελευταία στοιχεία της Eurocontrol για τις πτώσεις που δείχνουν αυτή τη διασύνδεση Ρουμανίας-Λιθουανίας μέσω της Αλβανίας. Αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Οπότε δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Αυτό ήθελα να σας πω, αγαπητέ συνάδελφε. Σας υπόσχομαι ότι θα προτείνω συμβαστικές τροπολογίες. Είμαι απόλυτα πρόθυμη και διαλεκτική να συζητήσουμε όλους τους συντάκτες των τροπολογιών και παρακαλώ διαβιβάστε ε, η βοηθή το μήνυμα προς τους ε, βουλευτές σας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το πόνιμά μας είναι σοβαρό για να ταράξουμε τα νερά και να κινηθούν τα πράγματα. με κυρία Φλότρ. Ο κύριος Έντσιο και πάλι. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, προσωπικός. Θα ήθελα να διατηρήσω την αξιοπρέπεια και το σεβασμό. Αλλά όταν μου λέτε ότι δεν είναι σοβαρή η πρότασή μου, θεωρώ ότι δεν είναι πολύ γενικό εκ μέρου τη κυρία Φλότρου. Κυρία Φλότρου, μα δεν είπα ότι δεν ήταν σοβαρό. Είπα ότι θέλω εξάπαντο να κάνουμε από κοινού μια σοβαρή δουλειά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. En tout cas, le point a été éclairé. πάντως, δεν είναι χαρακτηρισμός προσωπικό, αλλά πρόσκληση για σοβαρή δουλειά, για τη δουλειά που έχουμε ακόμη μπροστά μας. Τα έχουμε σχεδόν καταφέρει, τα έχουμε σχεδόν καταφέρει. Έχει τελειώσει και η ημέρα αυτή. Ευχαριστώ όλους και όλες σας που επιβιώσατε μέχρι τώρα και σας καλώ να τα ξαναπούμε στις 9 Ιουλίου στην προσεχή τακτική μας συνεδρίαση αν δεν απατώμε 9 και 10 Ιουλίου η προσοχή μας συνεδρίαση. Ευχαριστώ.